Τα έλεγα τα σήμερα και δεν με ακούγατε, τι κρίμα. Εντάξει, πάμε πάλι. Χαίρομαι λοιπόν που είναι τουλάχιστον 12 βουλευτέ εδώ σήμερα. Δεν μου αρκεί αυτό ο αριθμό, αλλά εν πάση περιπτώσει βάσει κανονισμού επαρκεί ο αριθμό. Αυτό περνάμε στην έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει, Όχι, ωραία. Περνάμε στο 2 τη ημερήσια διάταξη, τη ανακοινώσεις του Προέδρου η όμορφη αυτή συνεδρίαση θα μεταφερθεί στο στο ίντερνετ. Δεν έχουμε στονικά, λετωνιακά, λετωνικά, μαλτέζικα και σουηδικά. Ο κύριος Σούμπελ βρίσκεται εδώ για τελευταία φορά σήμερα μου ανέφεραν για τη μόνιμη είναι η μόνιμη σύνδεση, αν θέλετε, ο, μον, ο μόνιμος κρίκος μεταξύ ημών και της Επιτροπής. Είμαστε πάντα πολύ ικανοποιημένοι για τη συνεργασία που είχαμε. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Σούμπελ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σούμπελ ο οποίος φεύγει. Δεν συνταξιευωτείτε. Πάει στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Περνάμε τώρα στο 3 της ημερησίας διάταξης. Χαίρομαι που η Επίτροπος ε, είναι ήδη εδώ. Σας ε, καλωσορίζουμε, Ανδρούλα Βασιλείου. Πάει καιρός που σας είδαμε την περασμένη φορά. Οκτώ μήνες, αν δεν κάνω λάθος, ε, έχετε να έρθετε εδώ στην Επιτροπή μας. Τον Ιανουάριο ή ακούσαμε την κυρία Ρέντινγκ, τον Απρίλιο την κυρία Κλώσ. Χαιρόμαστε λοιπόν που ήρθατε σήμερα Είχε προγραμματιστεί άλλωστε η επίσκεψη, είχε ε, μάλλον προγραμματιστεί και άλλη επίσκεψη, αλλά είχε παρουσιαστεί μια δυσκολία εκ μέρου σα, οικογενειακό πρόβλημα στην Κύπρο και δεν μπορέσατε να έρθετε. Χαιρόμαστε που είστε εδώ πέρα όχι μόνο για να μας αναφέρετε τι θα κάνουμε σήμερα και το, του χρόνου, αλλά θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε και τα επόμενα πολιτή προγράμματα. Γιατί δεν μπορούν να μας πέσουν στο κεφάλι το Σεπτέμβριο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Υπάρχουν τόσε φήμες. Ξέρετε ότι στο τέλος οι φήμες γίνονται ολόκληρο τσουνάμι. Παίρνουν πολύ μεγάλες διαστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν αν θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγο την ευρύτερη εικόνα για το τι προγραμματίζει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τομέα της εκπαίδευσης, της ε, ε, ε του πολιτισμού. Ξέρω ότι θα υπάρξει σχετικό σχέδιο το καλοκαίρι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είμαστε διαθέσιμοι. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε λίγη παραπάνω σαφήνεια. Και φυσικά με την παρουσίασή σας θα σας θέσουν και οι συνάδελφοι ερωτήματα. Ελπίζω να είμαστε όλοι πάρα πολύ ευγενικοί και φιλικοί, γιατί όλα αυτά που θα μας πείτε ελπίζουμε να μας παρουσιάσετε πράγματα που θα μας διαβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ Επίτροπε και σας δίνω το λόγο. You have the floor. Uh, you, you want now? No. No, no, no, no. Ah, no. Okay. no it was first. <laughs> yes, yes, okay. Well, uh, dear Doris, uh, dear... Αγαπητοί Ντόρις, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι πάλι εδώ και όπως είπε και η Πρόεδρος πριν από λίγο, δυστυχώς δεν μπορούσα να έρθω την τελευταία φορά που προβλεπόταν κάτι τέτοιο, γιατί ένα δυσάρεστο γεγονός συνέβη στη χώρα μου. Ωστόσο πιστεύω ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή η συνεδρίασή μας αυτή. Τους τελευταίους μήνες η συνεργασία μας έχει οδηγήσει σε επιτυχίες με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Σήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πρόκειται, πιστεύω, για ένα πολύ καλό δείγμα δουλειά και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε στο πνεύμα αυτό. Την τον προηγούμενο μήνα στο Στρασβούργο, πολλοί συμμετείχαμε στην κοινή συζήτηση που έλαβε χώρα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η συζήτησή μα αποκάλυψε τελικά ότι έχουμε ένα κοινό όραμα για το τι είναι σημαντικό για του πολίτε μα και πού μπορεί τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τα πράγματα. Η παιδεία και ο πολιτισμός χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις αν πραγματικά, πρέπει, πραγματικά θέλουμε να δερματίσουν ένα πλήρη ρόλο στην κοινωνία. Σε στιγμές οικονομικής κρίσης πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στις πηγές της μελλοντικής ανάπτυξης. Αυτό ισχύει και για τη δουλειά που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκεί δηλαδή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να φέρει μια προστιθέμενη αξία στη δουλειά που, έρχεται, στη δουλειά που γίνεται στα κράτη-μέλη. Στο δεύτερο ήμιση του έτους θα προχωρήσω σε μια ανακοίνωση για τον εξυγχρονισμό της ανώτερης εκπαίδευσης. Πρόκειται για μία από τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 και για ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της στρατηγικής νεολαία κινήση. Ένας από τους στόχους μας για την Ευρώπη 2020 είναι, όπως το γνωρίζετε, ότι τουλάχιστον 40% από του νέου μα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πέρα από τα κοινωνικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα της ανώτατης εκπαίδευσης, θα βοηθήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την Ευρώπη να συμπληρώσει τα 16 εκατομμύρια, τις 16 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες απαιτούν ανώτατα προσόντα μέχρι το 2020. Δεν αρκεί όμως να έχουμε απλώς ένα ποσοτικό στόχο. Θα πρέπει να μας απασχολήσει και το είδος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο θέλουμε τα επόμενα χρόνια. Επομένως η ανακοίνωσή μου θα προσπαθήσει να ταποκριθεί σε κάποια δύσκολα ζητήματα. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα έχουν ε, ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Τι είδος σχέση θέλουμε να δημιουργήσουμε με τις επιχειρήσεις. Πώς θα βοηθήσουμε τα πανεπιστήμια μας να, ανοίξουν, να ανοιχτούν περισσότερο προς τον κόσμο και να καταφέρουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στο παγκόσμιο προσκήνιο. Πώς θα βοηθήσουμε τους φοιτητέ, τους διδάσκοντες και τους ερευνητέ να αναπτύξουν μεγαλύτερη κινητικότητα. Πώς θα καταφέρουμε να προωθήσουμε την δυνατότητα έβρεση εργασία για τους πτυχίουχους και πώ θα καταφέρουμε να προσπίσουμε την γνώση αυτή καθ' αυτή. Όλα αυτά τα ερωτήματα γίνονται ακόμα πιο επίγοντα τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττεται από μια βαθιά οικονομική κρίση. Βλέπουμε ότι ε, η ενεργεία των νέων έχει φτάσει το 40% σε ορισμένε χώρε και βλέπουμε ότι αυτό οδηγεί σε αισθήματα αγανάκτηση και οργή ανάμεσα σε μια, στους πολίτες μιας ολόκληρης Όταν οι νέοι αρχίζουν να χάνουν την ελπίδα στο μέλλον, αρχίζουν και αφισβητούν τελικά τις πιο τα πιο βασικά μας θεσμικά όργανα. Η ίδια η δημοκρατία μας τελικά διακυβεύεται. Θα πρέπει να δούμε τα φαινόμενα αυτά ως μια προειδοποίηση κινδύνου και ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράση συντομότατα. Πιστεύω λοιπόν ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να, αποτελέσει, να, να κατέχει μια νέα θέση στον προπολογισμό και την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο μέσω τη επένδυση και του εξοχρονισμού στα συστήματα τα εκπαιδευτικά μα θα καταφέρουμε να εξοπλίσουμε του πολίτε μα για μια κοινωνία που θα βασίζεται στην γνώση και που θα γίνεται όλο και πιο παγκόσμια. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε τις νέες αυτές δεξιότητες για τη νέα αυτή οικονομία και για μια πιο έντονη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει τις προτάσεις της για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν όμω τώρα η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για αριθμητικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει την τελική τη απόφαση στο τέλο του μήνα και αυτό θα γίνει από το κολέγιο όλων των επιτρόπων, προσπαθώντα να εξισορροπήσουμε τι διαφορετικέ μα αρμοδιότητε. Θέλω όμω να γνωρίζετε ότι εγώ χρησιμοποίησα όλη μου την ενέργεια, και αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία, αλλά πάλι οι συνεδριάσει έλαβαν χώρα με πάρα πολλού επιτρόπου, ιδιαίτερα με τον Επίτροπο για τον Προπολογισμό, με τον Πρόεδρο Μπαρόσο, Στην τελευταία μας ε, συνάντηση που έφερε τον, ε, την ονομασία εξομολογήσεις ε, ήταν παρόν και ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι και σε όλες αυτές λοιπόν τις συνεδριάσεις χρησιμοποίησα όλη μου την ενέργεια προκειμένου να ζητήσω μια σωστή κατάλληλη χρηματοδότηση για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει πολύ σημαντικούς στόχους στη στρατηγική 2020. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι για άλλη μια φορά. Ακόμα και σε μια περίοδο λιτοτητα μια πολιτισμένη κοινωνία θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει, να επενδύει στην εκπαίδευση, στην παιδεία των πολιτών τη. Στη σημερινή Ευρώπη ο λαό μα είναι η πηγή της μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι και εσεί θα με στηρίξετε στον δύσκολο αυτό αγώνα γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι για τα σημαντικά ζητήματα. Όλοι συνειδητοποιούμε ποια είναι η σημασία τη εκπαίδευση, τη παιδεία και του πολιτισμού σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Όλοι γνωρίζουμε ότι απαιτούν σημαντική δημόσια επένδυση και χωρί τι επενδύσει αυτέ δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε του στόχου Ευρώπη 2020. Όλοι θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερε ευκαιρίε κινητικότητα προκειμένου όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι όλων των ηλικιών να είναι σε θέση να σπουδάσουν, να διδάξουν και να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό. Όλοι πιστεύουμε στην αξία της διαβίου μάθησης. Αλλά θα ήθελα να είμαι σαφή. Αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, τότε χρειάζεται μια μεγαλύτερη επένδυση στην παιδεία και τον πολιτισμό, καλύτερη κινητικότητα των πολιτών μας και προκειμένου να επιτευχθούν αυτά δεν μπορούμε να παραμείνουμε στο εφιστάμενο status quo. Δεν μπορεί η κατάσταση να παραμείνει ως έχει από τους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι υπερασπίζονται τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Θεωρώ ότι αποτελούν μια επιτυχία και μπορούν να είμαστε περήφανοι. Με ένα χαμηλό κόστος πραγματικά αλλάζουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Και το όνομα Εράσμους πλέον αποτελεί ένα σύμβολο για τις ευκαιρίες που δίδονται και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οτιδήποτε και να κάνουμε στο μέλλον θα πρέπει να διατηρήσουμε τα καλά διδάγματα του παρελθόντος. Θα πρέπει όμως να είμαστε και ειλικρινεί κάθε φορά που συνειδητοποιούμε ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Τα τελευταία δύο χρόνια κάποια πολύ σημαντικά πράγματα έχουν όντω αλλάξει. Ακόμα αισθανόμαστε τι επιπτώσει τη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία ασκεί μια τεράστια πίεση στα δημόσια οικονομικά. Όλοι λοιπόν έχουμε καθήκον να δαπανούμε τα δημόσια χρήματα όσο πιο αποτελεσματικά και όσο πιο έξυπνα γίνεται. Και βλέπουμε βέβαια ότι η κρίση επιβαρύνει ιδιαίτερα τους νέους σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολλές φορές ε, απειλεί ακόμα και την κοινωνική ειρήνη. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οτιδήποτε και αν κάνουμε, οποιοδήποτε και ευρώ να δαπανούμε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να καταφέρουμε να βελτιώνουμε τους εαυτούς μας στο μέλλον στο υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο η υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεολαία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ιδιαίτερα κατακαιρματισμένη. Υπάρχουν πολλά και διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν διαφορετικού στόχου, καλύπτουν διαφορετικέ περιφέρειες του κόσμου, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και δεν υπάρχει, μάλλον η διασύνδεση μεταξύ του είναι αρκετά περιορισμένη. Είναι πολύ δύσκολο να αποτιμήσουμε αν τελικά η κατακαιρματισμένη αυτή κατάσταση εξυπηρετεί του μακροπρόθεσμου πολιτικού μα στόχου. Θα πρέπει να κρατήσουμε τα στοιχεία αυτά που λειτουργούν καλύτερα και θα πρέπει να καταφέρουμε να προωθούμε την κινητικότητα και τη διασυνοριακή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της εκπαίδευσης, είτε πρόκειται για μαθητές, είτε πρόκειται για φοιτητές, είτε πρόκειται για διδάσκοντες, καθηγητές, δασκάλους, εθελοντέ, ερευνητές. Μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο αυτό και παράλληλα μπορούμε να καταφέρουμε να απλοποιήσουμε τις δραστηριότητές μας προκειμένου να έχουμε μία ενιαία συνεκτική στρατηγική η οποία θα εξυπηρετεί τους στόχους ε, της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε το μελλοντικό μας πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την νεολαία σε τρεις βασικές δράσεις. Πρώτον, Κινητικότητα όσον αφορά την εκμάθηση. Στη συνέχεια, μεταρρύθμιση τη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ επίση και στι τρει χώρε, ιδίω όσον αφορά τον εξυγχρονισμό τη ανώτατη εκπαίδευση. Και τέλο, συνεργασία και καλύτερε εταιρικέ σχέσει μεταξύ των εκπαιδευτικών Ινστιτούτων και των άλλων ενδιαφερομένων. Για παράδειγμα, ένα πιο ενισχυμένο διάλογο ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τι επιχειρήσει. Οι τρει αυτέ δράσει αλλοσυμπληρώνονται. Ενδυναμώνει μία την άλλη. Προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικέ, θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα ενιαίο πρόγραμμα με όλα τα ωφέλη που αυτό μπορεί να αποφέρει. Ένα τέτοιο ενιαίο πρόγραμμα θα εξασφαλίσει το οτιδήποτε κάνουμε τελικά συμβάλλει στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η εκπαιδευτική μα στόχη, ο εξυγχρονισμό των τη εκπαίδευση, καθώ επίση και η στρατηγική μα για την νεολαία. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουν λιγότερε και πιο απλέ διαδικασίε και οι διαχειριστέ των προγραμμάτων θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν πιο απλά και ξεκάθαρα εργαλεία. Η ταυτότητα των προγραμμάτων, των προγραμμάτων μας, το προφίλ των προγραμμάτων μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ονόματα όμως, οι λογότυποι, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καθορίσουν την πολιτική μας. Καταρχάς θα πρέπει να καταλήξουμε στη σωστή πολιτική και μετά να αποφασίσουμε ποιο θα πρέπει να είναι το σωστό όνομα της πολιτικής αυτής. Θα ήθελα τέλος να σας ενημερώσω για κάποιες σκέψεις που κάνουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο στα πλαίσια των νέων προγραμμάτων μας. Σήμερα υπάρχουν όλο και περισσότεροι νέοι οι οποίοι σπουδάζουν, προσπαθούν να κάνουν ένα μάστερ και δεν έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Ελάχιστε είναι οι χώρε αυτέ που προβλέπουν δανειοδότηση φοιτητών προκειμένου αυτοί να σπουδάσουν σε μια άλλη χώρα και θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί με το παραδοσιακό πρόγραμμα Εράσμους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που κάνουν μάστερ. Θα ήθελα να καλύψω λοιπόν το κενό αυτό δημιουργώντας ένα πρόγραμμα εγγύησης το οποίο θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνονται εθνικέ τράπεζε Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνουν δάνεια προς φοιτητές. Κατά αυτόν τον τρόπο χιλιάδε παιδιά θα καταφέρουν να σπουδάσουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα μάστερ στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας από την οποία προέρχονται. Θα ήθελα βέβαια να τονίσω ότι το σύστημα αυτό παροχής εγγύσεων θα έρθει να προσθεθεί στο εφιστάμενο σύστημα επιδοτήσεων που έχουμε για την πρόθεση της κινητικότητας. Η, πρόθεση, η καινοτόμο αυτή προσέγγιση για τη χρηματοδότηση, καθώ επίση και η γενικότερη πρόθεση να πλουστεύσουμε τα προγράμματά μα, ουσιαστικά συνάδει με τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε ζητήσει στο παρελθόν να γίνουν αυτέ οι μεταρρυθμίσει. Θα ήθελα να περάσω τώρα στον τομέα του πολιτισμού. Προφανώ μα έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και το μέλλον του ε, των προγραμμάτων μα για τον πολιτισμό και τα προγράμματα media. Θα ήθελα να αναπτύξω και τα δύο αυτά προγράμματα και θα ήθελα να εξασφαλίσω την αυτονομία τους, καθώς επίσης ότι θα χαίρουν της κατάλληλης χρηματοδότησης. Έχουμε συζητήσει εκτενώς την αξία των προγραμμάτων αυτών και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την υποστήριξή σας. Συζητήσαμε και για το πώς θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κλάδο του πολιτισμού και των καινοτόμων ε, βιομηχανιών, αν θέλετε, δραστηριοτήτων μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να εντάξουμε καλύτερα τον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική το 2020 και θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για τον πολιτισμό η βιομηχανία, θέλετε, του πολιτισμού, το, τομέα του πολιτισμού αντιστοιχεί στο 4,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Υπάρχουν όμω κάποια διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι περισσότερε επιχειρήσει λειτουργούν σε μια αγορά η οποία είναι ιδιαίτερα κατακαιρματισμένη και δεν έχουν την απαραίτητη δεν έχουν τι απαραίτητε επενδύσει. Επίση, δεν καταφέρνουν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχουν μάλλον έχουν πάντα μια βέβαιη εμπορική επιτυχία οι περισσότερε από αυτέ τι πολιτιστικέ επιχειρήσει και δεν έχουν και εξασφαλισμένη πρόσβαση σε δενεδότηση από τι τράπεζε. Εδώ, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε εμεί να αλλάξουμε τα πράγματα. Έχω αρχίσει να εξετάζω ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο θα δίδει εγγυήσει στι τράπεζες και με τη συνέχεια οι τράπεζες θα μπορούν να δανειοδοτούν κάποιες εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να δίνουν και στις επιχειρήσεις ένα πρώτο κεφάλαιο εργασίας. Υποστηρίζω λοιπόν την ιδέα αυτή γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα ενθαρρύνει τις τράπεζες να ενισχύουν περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπορούν επίσης να καλύπτουν κάποια στοιχεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα, πνευματικά δικαιώματα. Επίσης πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κάποιες οικονομίες κλίμακος μέσω του, μέσω του συστήματος αυτού, προκειμένου να βοηθήσουμε τις μικρές αυτές επιχειρήσεις και θα καταφέρουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την ίδια θετική εμπειρία που υπάρχει από κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το υπόλοιπο των κρατών μελών. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για τον αθλητισμό. Πιστεύω πραγματικά ότι ο αθλητισμό θα πρέπει να έχει μια ξεχωριστή θέση στον κοινοτικό προπολογισμό και αυτό παραμένει ο στόχο μου. Όλοι γνωρίζουμε ποιε είναι οι δημοσιονομικέ πιέσει εκείνε οι οποίε έχουν περιορίσει την κοινοτική δράση στον τομέα αυτό. Οι πιέσει αυτέ προφανώ δεν έχουν εξαφανιστεί Πιστεύω πάντως ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για τον αθλητισμό, το οποίο θα αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές προκλήσεις που εμφανίζονται στον τομέα του πολιτισμού και που θα προωθεί την κοινωνική και εκπαιδευτική πτυχή του αθλητισμού. Όλο και περισσότερο σήμερα βλέπουμε ότι η διαχείριση του αθλητισμού, το του αθλητισμού θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο υποστηρίζοντα ομοσπονδίε εκείνε αθλητικέ οι οποίε θέλουν να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργία του. Μέσα στον χρόνο αυτό θα έχουμε και μία συνδιάσκεψη η οποία θα επικεντρωθεί στο ζήτημα αυτό και θα αποτελέσει συνέχεια της έντονης συζήτησης που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα αποτελέσει συνέχεια και της μελέτης που δημοσιοποίησε λίγο νωρίτερα φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα Ήθελα επίσης να ενθαρρύνω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταφέρουν να καταπολεμήσουν τα παράνομα στοιχήματα και γενικότερα την νοθεία και την απάτη στον αθλητισμό. Καταλαβαίνετε ότι προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει ένας κοινοτικό συντονισμό, συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αγαπητοί συνάδελφοι, προκειμένου να τα πετύχω όλα αυτά χρειάζομαι την δική σας υποστήριξη. Σίγουρα μας περιμένει μια πολύ δύσκολη μάχη. Όχι μόνο με στα θεσμικά όργανα, αλλά και με κάποια άλλα συμφέροντα ή ακόμα και με ένα τμήμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πιστεύω πάντως ότι τα επιχείρηματά μας είναι βάσιμα και πιστεύω πραγματικά ότι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν μια ξεχωριστή χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προπολογισμό εφόσον με χαμηλό κόστος αποφέρουν τεράστια ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες αν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και πιστεύω ότι συμφωνούμε για κάποιε πολιτικέ προτεραιότητε, τότε θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μαζί έναν προπολογισμό που θα δώσει νέε δυνατότητε, νέε ευκαιρίε στου πολίτε μα. Ένα προπολογισμό που θα βοηθήσει του πολίτε μα να πετύχουν ε, το απόλυτο δυναμικό του ε, σε μια μελλοντική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you. I was very attentive. Σα ευχαριστούμε, Ανδρούλα. Με πολύ προσοχή σας άκουσα και ε, προσέλαβα το μήνυμά σας. Ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα, είπατε. Όχι εκπαίδευση, νεολαία και προγράμματα στον πληθυντικό. Όχι, πρόγραμμα στον ελληνικό. Είναι σαφές. Αυτό που θέλαμε να αποφύγουμε πριν από 1,5 χρόνο τώρα μας χτυπάει πίσω πισόπλατα. Δεν είμαι μόνιμο τόσο στη συζήτηση αυτή. Πολλές ε, εισηγήσει. Ε, πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο για να θέσουν ερωτήσεις. 11, 12, 13. Α, και κλείνει ο κατάλογος. Τελευταία κυρία Κώστα και κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. να σας ζητήσω να είστε πάρα πολύ σύντομοι, να μην κάνετε γενικά σχόλια. Δύο λεπτά. Μάξιμουμ. Η κυρία Παντία. Μένος de dos minutos porque... Θα χρειαστώ λιγότερο από δύο λεπτά. Απλά θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να πάω στην Επιτροπή Βιομηχανία επειδή υπάρχει μια γνωμοδότηση ακριβώ για το θέμα νέε δεξιότητε, νέε θέσει εργασία. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τι ε, πολύ λεπτομεριακέ επεξηγήσει που μα έδωσε. Δυστυχώ δεν μπορώ να παραστώ. Υπάρχουν πολλέ ερωτήσει. Είμαι πεπισμένη ότι θα διατυπωθούν τα ερωτήματα που θα με ενδιέφεραν και βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον ε, θα ενημερωθώ για τι απαντήσει και ζητώ συγγνώμη για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα ενημερώσετε και την ε, συντονιστριά σας, την κυρία Χανιμπάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, γιατί και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο, δεν μιλάω για τον προπολογισμό τώρα, γιατί το θέμα αυτό θα το εξετάσουμε στη συνέχεια και ξέρω ότι η, επίτροπο Επίτροπος ε, θέλει να δώσει σκληρό αγώνα για να πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά για να καταλάβουμε κάτι παραπάνω, θα υπήρξε δηλαδή ένα ενιαίο πρόγραμμα για την κινητικότητα, για την εκπαίδευση. Και θα διατηρηθεί το πρόγραμμα για τον πολιτισμό, θα υπάρχει το πρόγραμμα για τα μέσα και ένα τέταρτο πρόγραμμα για τον αθλητισμό και θα συμπεριληφθεί στη συνέχεια ο αθλητισμός και στα τρία αυτά προγράμματα. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις για τα μεμονωμένα προγράμματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υπάρξει κάποιο πλαίσιο. Και όταν θα υπάρξουν ενδεχομένω οι ανακοινώσεις αυτές. Θα ήθελα να υπολογίζω πότε, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις για να είμαστε σαφείς, για να μην ρωτάμε τρεις φορές τα ίδια πράγματα, λέει η Πρόεδρος. Η Επίτροπος μας ενημέρωσε εκ των προτέρων σχετικά με αυτά που θα μας ανακοινωθούν επίσημα μετά τις 29, δηλαδή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο. Μας εξήγησε η Επίτροπος ότι ήδη θα υπάρξει ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την νεολαία, καταρχάς ένα πρόγραμμα πολιτισμού και για τα μέσα και ελπίζει να υπάρξει και ένα πρόγραμμα για τον αθλητισμό. Αυτή η ελπίδα μου φαίνεται κάπως φιλοδόξη. Να εξηγήσουμε λοιπόν πώ έχει η κατάσταση για να μην θέτουμε συνέχεια τι ίδιε ερωτήσει. Πρόκειται για μια πρώτερη ενημέρωση ε, σήμερα. Η πραγματική ενημέρωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρθει μετά τι 29 Ιουνίου. Θα έχουμε λάβει τα στοιχεία αυτά πλέον εγγράφω και θα δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε τότε. Ο κύριο Μπάγκο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κυρία Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαιτέρως ε, που ήρθατε ξανά στην Επιτροπή μας. Δύο σύντομα ερωτήματα έχω να σας απευθύνω. Το πρώτον, πώς νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με αναπηρίες να συμμετέχουν περισσότερο, να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή γενικώς. Και επίσης, θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα μπορούσαμε να, τα, ε, να τους δώσουμε μια καλύτερη πρόσβαση. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τον αθλητισμό, υπήρξε αυτή η πρόταση για ένα πρόγραμμα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε σαν Επιτροπή να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Φυσικά δεν θα σας εκπλήξω ότι θα μιλήσω και εγώ για τον αθλητισμό. Υπήρξατε επίτροπος ε, αρμόδια για την υγεία νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και γνωρίζετε επίσης ότι η προαγωγή του αθλητισμού μπορεί να φέρει εξοικονομήσεις, οικονομίες στον τομέα της υγείας. Δηλαδή η σωματική δραστηριότητα, η αθλησή μπορεί να έχει ωφέλη και στον τομέα της υγείας. Άρα και αυτός θα μπορούσε να είναι ένας λόγος υπέρ της χρηματοδότησης του αθλητισμού. Εσείς σας ε, επισημάνατε τη σημασία του προγράμματος Εράσμους ή μάλλον των προγραμμάτων Εράσμους. Νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν γιατί ε, νομίζω ότι το Εράσμους έχει κάνει πολύ περισσότερα από πολλές συνθήκες για τους Ευρωπαίους και το Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλδημοκράτες, ε, ίσω θα υπάρξει και στήριξη από του ελευθέρους. Εμεί λοιπόν οι τρει τα τρεις πολιτικέ ομάδε, θα θέλαμε να κάνουμε μια πρόταση για ένα πιλωτικό πρόγραμμα τύπου Εράσμου για τον αθλητισμό. Επίση θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο και το θέμα τη κινητικότητα που αναφέρατε. Ξέρετε ότι υπήρξε στην Ισπανία ένα μεγάλο κίνημα και σε άλλε χώρε, η αγανακτισμένη λέγεται αυτό το κίνημα, ε, πάρα πολλοί άνεργοι, πάνω από το 45% αποφύτων πανεπιστημίου στην Ισπανία είναι άνεργοι. Καταλαβαίνω ποια είναι τα προβλήματα, ε, τα κατανοώ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε τις πανεπιστημιακές σπουδέ να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες της αγοράς. Αφενός. Αφετέρου πρέπει να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε την επαγγελματική εκπαίδευση που πάντοτε θεωρείται δευτέρας κατηγορίας. Και θα έλεγα και την εκμάθηση γλωσσών Καλή είναι η κινητικότητα, ε, αλλά αν κάποιος θέλει να εργαστεί στη Γερμανία ή στην Ελλάδα θα πρέπει να ξέρει ελληνικά, γερμανικά. Άρα πρέπει να γίνει προσπάθεια για την εκμάθηση γλωσσών. Έτσι θα πετύχουμε νομίζω την κινητικότητα και θα αποφύγουμε και την νεανική ανεργία. Ευχαριστώ. Ε, για τα θέματα του ενιαίου προγράμματος για την νεολαία και για τον πολιτισμό. Μία ερώτηση. Πώς ε, θα διασφαλίσετε ότι όλα αυτά θα μπουν ε, σε ένα πρόγραμμα και έτσι θα αντικατασταθούν στο μέλλον και τα επιτυχημένα προγράμματα του παρελθόντος. Πώς θα διαμορφωθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, πώς θα διασφαλίσετε αυτή την επιτυχία, τι θα γίνει στο ιστορικό του προγράμματος, ποια θα είναι η διάρθρωση δεδομένου ότι σε κάθε χώρα είναι διαφορετικές οι ανάγκες που υπάρχουν. Τι θα γίνει και με την προώθηση της επαγγελματική κατάρτισης. Και έχω υπόψη μου την επιτυχία του Λεωνάρδο Νταβίντσι, του Εράσμους, του Κομένιους, η οποία, τα οποία καθιέρωσαν την κινητικότητα. Θα συνεχιστούν όλα αυτά σε ένα ενιαίο πρόγραμμα και πώς θα διασφαλίσετε όταν θα υπάρχει ένα πρόγραμμα στα οποία θα συνενωθούν όλα αυτά τα στοιχεία πώς θα επαρκέσει για τον όλο ένα και πιο περιορισμένο προϋπολογισμό. Πώς θέλετε να διασφαλίσετε αυτά που είπατε, η ενίσχυση, η επέκταση, η μεγαλύτερη ενίσχυση της ε, παιδείας στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. Πώς θέλετε λοιπόν να διασφαλίσετε ότι όλα αυτά θα διατηρηθούν στη συνένωση σε ένα πρόγραμμα. Και... Ε, ε, Ευχαριστώ τελευταία η κυρία Τρίπελ, η αντιπρόεδρος κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω ότι ο στόχος της Επιτροπής Βασιλείου, ότι τα μέσα για τα προγράμματα πολιτισμού και για όλες τις υπόλοιπες αρμοδιότητάς μας με βρίσκουν σύμφωνοι. Και θεωρώ ότι η στρατηγική για το 2020 έχει ως δοδηλωμένο στόχο να αφιερώσει πιο πολλά για την έρευνα, την ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την πολιτισμική ποικιλία και το καθεξής. Αλλά θα ήθελα και είχαμε και προηγουμένως την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, να επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Φερχάιεν. Αν λόγω τακτικών ε, λόγων θέλουμε να αλλάξουμε την ονομασία και να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα ομπρέλα μήπως ε, στις δύσκολες εποχές που ζούμε υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε πιο πολλά από ό,τι θα κερδίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ακούσω, κυρία Επίτροπε, την ακριβή στρατηγική σας. Πώς σκοπεύετε να τα διασφαλίσετε αυτά για να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή. Γιατί μόνο τότε θεωρώ ότι θα σας υποστήριζε η Επιτροπή Πολιτισμού. Αν δεν πιστούμε, γι' αυτό θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Uh, Καταρχάς θα σας μιλήσω λίγο για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Όπως είπα στα τέλη του τρέχοντος μηνός θα εγκρίνουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα θα αποφασίσουμε για τον προϋπολογισμό και τις διάφορες κατηγορίες του. Τόσα για την εκπαίδευση, τόσα για τον πολιτισμό κτλ. κτλ. Και τότε θα ληφθούν και θα ολοκληρωθούν, θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για την αρχιτεκτονική των προγραμμάτων μας. Μάλλον κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα γίνει αυτό. Μόνο τότε η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων και οι δικές μας προτάσεις για τα προγράμματα θα εγκριθούν τότε. Επομένως, την περίοδο που θα μεσολαβήσει μέχρι την έγκριξη θα την εκμεταλλευτούμε, γιατί βέβαια καλό είναι να γνωρίζουμε τι προπολογισμό θα έχουμε διαθέσιμο για να διατυπώσουμε τι προτάσει μα για την αρχιτεκτονική των προγραμμάτων. Θα τον εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό το χρόνο. Αλλά είχα την εξή επιλογή. Από παντού υπάρχουν κλήσει για απλούστευση, για περικοπή, για μείωση του διοικητικού άχθου, για δημιουργία συνεργασία με τα διάφορα δημοσιονομικά εργαλεία. Μιλάω πάντα για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν γίνει αυτό, αισιοδοξώ, βέβαια δεν μπορώ να είμαι βέβαια, αλλά αισιοδοξώ, με βάση τις συζητήσεις που είχα, ότι θα μπορέσω να εξασφαλίσω αύξηση της χρηματοδότησης για τα προγράμματά μας. Αυτή είναι η προτεραιότητά μου. Διότι καμία από τις κατηγορίες δικαιούχων που σήμερα συμμετέχουν στα προγράμματα κινητικότητας δεν πρόκειται να φυγεί. Θα διατηρήσουν όλοι το δικαίωμα που έχουν προς κινητικότητα, είτε είναι θελοντές, είτε είναι νέοι που συνεργάζονται με άλλους νέους από άλλες χώρες, είτε είναι φοιτητέ, σπουδαστέ, εκπαιδευτικοί και ούτω καθεξής. Θα διατηρήσουν όλοι το δικαίωμα κινητικότητας όπως ισχύει μέχρι τώρα. Αλλά η πρόθεσή μου είναι να δείξω ότι ναι, αφενός Μπορούμε να περιστύλουμε το διοικητικό άχθος και γνωρίζετε από τις μελέτες που έχουν γίνει ότι κάποια προγράμματα ίσως είναι πολύ μικρής κλίμακας ώστε να μπορούν να έχουν κάποιο αντίκτυπο ή δεν έδειξαν ότι έχουν την προστιθέμενη αξία που θα αναμενόταν. Προσπαθώ λοιπόν να δω πώς μπορώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να είμαι πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική και βέβαια να φροντίσω τα προγράμματά μας να έχουν μεγαλύτερη προβολή, μεγαλύτερη ορατότητα. Αυτή ήταν η επιλογή που είχα και αυτό επέλεξα. Δεν έχω αποφασίσει ακριβώς πώς θα ονομάσω ε, το πρόγραμμα, πώς θα το σχηματίσω, πώς θα το διαμορφώσω, αλλά η φιλοσοφία είναι αυτή που σας αναφέρω. Βέβαια, όπως είπε και η Ντόρις, έχουμε ένα πρόγραμμα για την παιδεία, την εκπαίδευση δηλαδή την, ε, και την επαγγελματική κατάρτιση και την νεότητα, αλλά θα έχει διάφορα σκέλη για τους εκπαιδευτικούς, για τους ειδητές, ε, για τους εθελοντές κτλ. Θα λάβουμε επίσης υπόψη τη διεθνή πτυχή των προγραμμάτων αυτών, διότι σήμερα έχουμε το Erasmus Mundus ως ξεχωριστό πρόγραμμα. Θέλουμε να το εντάξουμε και αυτό στο πρόγραμμά μας. Και έπειτα θα έχουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα πλαίσιο για τον πολιτισμό, αλλά με μεμονωμένες συνιστώσεις. Πολιτισμός, μήμη και αν έχουμε κάποια επιπλέον κονδύλια, αυτό που σας είπα, παιδεία και δημιουργική βιομηχ... δημιουργικές βιομηχανίες. Αλλά το πρόγραμμα, τα προγράμματα μάλλον για τα ΜΜΕ και για την παιδεία θα είναι διαφορετικά, θα είναι αυτόνομα και θα έχουν το δικό τους προπολογισμό. Και στόχος δικός μου αλλά και του κυρίου Λεβαντόφσκι ήταν να υπάρξει και ξεχωριστό πρόγραμμα για τον αθλητισμό. Ίσως να μην είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα, αλλά θέλουμε να υπάρχει παρόλα αυτά ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για τον αθλητισμό. Τους μίλησα για τις διάφορες δράσεις που θέλουμε να αναλάβουμε και οι οποίες δεν έχουν να κάνουν τίποτα ούτε με την παιδεία ούτε με τον πολιτισμό. Παραδείγματο χάρη, ε, η δυτή εκπαίδευση, το dual training, ναι, μπορεί να έχει κάτι να κάνει και με την εκπαίδευση, αλλά οι περισσότερες άλλες δράσεις δεν έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Είπα λοιπόν ότι δεν θα έπρεπε να θυσιάσουμε ένα πάρα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα για να εξοικονομήσουμε δεν ξέρω κι εγώ πια πόσα εκατομμύρια που είναι ψίχουλα σε σχέση με το συνολικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά έχω κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να το πετύχω αυτό. Μετέφθη ένα ιδιαίτερο, ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τα άτομα με αναπηρία. Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι να δώσουμε ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Όταν μιλάω για ισότητα, μιλάω για όλα τα παιδιά. Είτε έχουν μια σωματική αναπηρία, είτε διανοητική, είτε προέρχονται από φτωχό περιβάλλον, σε μειονεκτική θέση. Ε, θέλουμε να του δώσουμε σε όλα αυτά τα παιδιά τις ίδιες δυνατότητες. Δεν έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά με αναπηρία, γιατί αυτό εντάσσεται στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών. Στόχος μας όμως είναι να κατανοήσουν τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε όλα αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Τώρα, οι εγκάρσεις δεξιότητες για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάμε εδώ για την ανεργία και ιδίως για τους ανέργους νεαρούς αποφύτους. Γνωρίζετε ότι ακόμη και σήμερα που έχουμε 5 εκατομμύρια νεαρούς ανέργους, ακόμη και σήμερα εξακολουθούμε να έχουμε πολλές κενές θέσεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν διότι δεν βρίσκονται οι απαιτούμενε δεξιότητε. Μιλάμε για εγκάσει δεξιότητε, εκμάθηση γλωσσών, μιλήσατε για τι γλώσσε. Λήψη αποφάσεων, ομαδική εργασία, προσαρμοστικότητα. Μπορεί κάποιο να σπουδάσει σε ένα αντικείμενο, αλλά να χρειαστεί να εργαστεί σε έναν εντελώ διαφορετικό τομέα. Θα πρέπει όμω να είναι κάποιο στη θέση να προσαρμόζεται στι νέε περιστάσει, στι νέε συνθήκε. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εγκάραση αδεξιότητα. Και αυτέ οι δεξιότητε νομίζω ότι είναι αυτέ που θα αποκτήσουν οι νέοι με την κινητικότητα. Γι' αυτό και θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην κινητικότητα Γι' αυτό και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να απαλείψουν όλους τους φραγμούς που εμποδίζουν την κινητικότητα. Παραδείγματο χάρη η μεταφορά των υποτροφιών ή των δανείων, μια αναγνώριση κάποιων επαγγελματικών προσόντων ή κάποιων μαθημάτων που κάποιος έχει περάσει σε ένα πανεπιστήμιο και δεν αναγνωρίζονται σε ένα άλλο και ούτω καθεξής. Ξέρετε επίσης ότι θα υπάρξει και ένα ετήσιο scoreboard για την κινητικότητα και θα βλέπουμε εκεί τις επιδόσεις όλων των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Και μετά θα βλέπουμε και θα προσπαθούμε να δούμε γιατί δεν μπόρεσαν κάποιες χώρες συγκεκριμένε να αυξήσουν την κινητικότητα των φοιτητών τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια εμπόδια υφίστανται και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να υπερπηδήσουν τις δυσκολίες αυτές που αντιμετωπίζουν οι νέοι τους. Νομίζω ότι έχω απαντήσει. Μάλιστα, μπορούμε να ακούσουμε τις επόμενες ερωτήσεις. Ο κύριος Λόκκαρτ. Øh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα πολλά να πω, αλλά η Επίτροπος απάντησε ήδη σε πολλές από τις ερωτήσεις. Ε, μία μικρή ερώτηση λοιπόν από πλευρά μου. Συμφωνώ με το όραμά σας. Θεωρώ όντω ότι είναι ορθό να ακολουθήσουμε την ιδέα αυτή και θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γεννηθούμε. Αλλά να ρωτήσω την Επίτροπο. Ξέρετε ότι ο κόσμος ανησυχεί για τα προγράμματα αυτά και ότι ανησυχεί για το τι θα συμβεί. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να δώσετε εγγυήσεις φυσικά, αλλά υπάρχει λίγο η ιδέα ότι ίσως κάποιοι, κάποια άτομα αμ, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν πιστεύετε ότι κάποιοι επιτρόποι υποστηρίζουν αυτές τις ιδέες. Τι γίνεται με το πρόγραμμα για τον αθλητισμό, για παράδειγμα, γιατί εδώ όλοι συμφωνούμε ότι όσο και όμορφα να ακούγονται τα προγράμματά σας, είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ο αθλητισμός. Και ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η διάθεση που επικρατεί μεταξύ των επιτρόπων. Σας ευχαριστώ. Ja vielen Dank. κυρία ευχαριστώ Επίτροπε, σας ευχαριστώ και για τις εξηγήσεις σας. Ήδη στην προηγούμενη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας, μας ανακοινώσατε ότι ως ε, Επιτροπή Πολιτισμού Μάλλον σα είπαμε ότι ω Επιτροπή Πολιτισμού θα είμαστε αντίθετοι σε ένα ενιαίο πρόγραμμα. Βλέπω ότι δεν αλλάξατε στάση. Και δεν έχω πιστεί ακόμα ότι αυτό αποτελεί μια σωστή και ορθή λύση. Να τα βάλουμε όλα σε ένα καλάθι, γιατί ίσως ε, έτσι θα ε, διακινδυνεύσουμε πράγματα τα οποία έχουμε αγαπήσει και έχουν μια παράδοση στην Ευρώπη. Μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είχαμε το πρόγραμμα Youth in Action, νεολαία σε δράση, σε ό,τι αφορά τη μη τυπική, μη επίσημη ε, εκμάθηση. Αυτό ήταν κάτι που μας απασχολούσε πάρα πολύ. Δεν θέλαμε μόνο την επίσημη εκπαίδευση, θέλαμε να συμπεριλάβουμε αυτά που κάνουν οι νέοι ε, στον ελεύθερο χρόνο τους, αυτά που μαθαίνουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Και ανησυχούμε λοιπόν ότι πλέον ο τομέας αυτός της ε, μη επίσημης εκμάθησης από το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση θα χαθεί λίγο, αν θέλετε, στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης. Και αυτό δεν θα μας έβρισκε καθόλου σύμφωνο ως Επιτροπή. Right. Έχετε δίκιο. Η κυρία σας ευχαριστώ, Επίτροπε, για τα σχόλια που κάνατε. Κοιτάξτε, σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ε, καθόλου περιορισμοί στον προπολογισμό και θα έπρεπε να μπορούμε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση όσο θέλουμε. Πρέπει όμως να δούμε πώς έχει τρέχουσα οικονομική κατάσταση και δεν μπορούμε να ζητούμε αύξηση στον προπολογισμό χωρίς να γίνει απολογισμό των επενδύσεων που γίνονται. Γι' αυτό συμφωνώ ότι πρέπει να δούμε τι λειτουργεί και τι όχι και είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα των επενδύσεων που κάνουμε στα προγράμματα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όντως πετυχαίνουμε ωφέλη, πλεονεκτήματα και προστιθέμενη αξία. Αναφερθήκατε στην εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση Εμένα αυτό που με περισσότερο είναι τα άτομα που βρίσκονται στο ενδιάμεσο διάστημα, δηλαδή όσοι έχουν φύγει από το σχολείο αλλά δεν καταφέρουν να πάνε στο πανεπιστήμιο. Τι μπορούμε να κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια των επιχειρήσεων θα, μπορέσα, θα μπορούσαμε να δώσουμε στους ανθρώπου αυτού να μάθουν στα πλαίσια των επιχειρήσεων ασκώντα μια δουλειά κάποια πράγματα. Και όσον αφορά τα προγράμματα media, Μήπως θα μπορούσαμε να βάλουμε στα προγράμματα αυτά και τη συνιστόσα όσον αφορά τα παιχνίδια στους υπολογιστές computer gaming. Όσον αφορά τώρα τον αθλητισμό, θα ήθελα να αφαιρθούμε και στον εθελοντισμό. Ξέρετε ότι ε, αυτή τη στιγμή γίνεται μία αναθεώρηση του τμήματος του τομέα αυτού και προβλέπονται για τον αθλητισμό τουλάχιστον κάποιες απαλλαγές και εξαιρέσεις από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Θα συνεχίσετε και εσείς να υποστηρίζετε αυτές τις φοροαπαλλαγές. Μην ε, υπερβαίνετε το χρονομιλία σας. Η κυρία Μποσκούρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω για τον αθλητισμό. Είμαι η συγγήτρια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και εξετάζω δηλαδή την πλευρά των ε, δικαιωμάτων των πολιτών. Αναφέρεται κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία για τους ε, διαμεσολαβητές ε, στον αθλητισμό και για το συνέδριο που θα διοργανωθεί, αλλά ανακοινώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά από πλευρά νομοθεσία. Τι θα προκύψει από την συνέδριο δηλαδή για τα νόμιμα στοιχήματα. Υπάρχει συμφωνία FIFA και Interpol. Αυτό μας επηρεάζει πάρα πολύ και στην Ευρώπη. Εσείς οι συνάδελφοί σας έχετε επαφές στο επίπεδο αυτό για να διεξαχθούν πανευρωπαϊκές ενέργειες και δράσεις. Και τελευταία ερώτηση. Αναφέρατε φυσικά ότι ο αθλητισμός αγγίζει όλους τους τομείς Υπάρχουν κάποια πολύ καλά προγράμματα συμφιλίασης όπου τα παιδιά ε, που παλιότερα ήταν ε, ε, το ένα αντίθετο με το άλλο και μάχονταν το ένα με το άλλο πλέον μπορούν να συμφιλιωθούν μέσω του αθλητισμού. Για την σταθεροποίηση των Βαλκανίων είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρω ότι είναι πολύ περιορισμένο ο προπολογισμό, αλλά μήπω θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον προπολογισμό για τι εξωτερικέ υποθέσει. Γιατί εγώ βλέπω πολύ σαφή πλέον εκτίματα και φαντάζομαι ότι και εσεί συμφωνείτε. Η πρόεδρο, ε, για τον επόμενο. Για το τρέχον έτος έχουμε συμπεριλάβει ε, τέτοια προγράμματα που ακριβώς αυτό το στόχο επιδιώκουν που ανέφερε η Έμιλη Μποσκούρτη. Κυρία Πελιοδέλη. Ε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα κυρία Βασιλείου να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και χαίρομαι ιδιαίτερα, περιμένω μάλιστα να δω σύντομα την αρχιτεκτονική της ε, χρηματοδότησης των προγραμμάτων. Ε, πιστεύω ότι μια εκλογήκευση όπως τη σκέφτεστε θα ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο γιατί μοιάζει τα προγράμματα και η χρηματοδότηση να είναι διάσπαρτα σε επιμέρους κατηγορίες. Ε, μια ερώτηση που αφορά στον εξυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης των πανεπιστημίων μας. Ε, αν κατάλαβα καλά, αντιλαμβάνεστε την εκπαίδευση ε, ως ε, ανεξάρτητη, όχι αναγκαστικά δεμένη με την επαγγελματική αποκατάσταση Μιλήσατε για learning in its own sake. Από την άποψη αυτή πώς σκέφτεστε να συμπεριλάβετε τις ανθρωπιστικές σπουδέ, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με τις ε, επιχειρήσεις ε, στον τρόπο με τον οποίο ε, σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό. Πώς μπορούν να ενταχθούν οι ανθρωπιστικές σπουδέ στον εξυγχρονισμό που για μένα είναι πολύ σημαντικό και μια ερώτηση που πάει παράλληλα θεωρείτε ότι με τον όρο έρευνα που αναφέρεστε στο κειμενάκι που διάβασα θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και η έρευνα των ανθρωπιστικών σπουδών γιατί είναι πραγματικά απογοητευτικό και το λέω από την προσωπική μου μεγάλη πείρα ότι με τον όρο αυτό συνήθως μιλούμε για research σε εργαστήρια ε, θετικών επιστημών. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να προβλεφθούν προγράμματα που να υποστηρίζουν και την πολιτιστική έρευνα. Αρχαιολογία, φιλολογία, ιστορία κλπ. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη στην αρχιτεκτονική ε, που ετοιμάζετε. Σας ευχαριστούμε. Πάνω. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ο δωδέκατος που θα θέσει την ερώτηση αυτή μάλλον που θα μιλήσει και πολλά ζητήματα ακούσαμε ήδη. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τους στόχους που μας παρουσίασε και οι οποίοι πραγματικά αξίζουν να τους υποστηρίξουμε. Και μιλώντα για τα προγράμματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η οικονομική, η χρηματοοικονομική πραγματικότητα πλέον έχει γίνει πιο σφιχτή Άρα τα χρήματα που έχουμε θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για τα πιο σημαντικά στοιχεία για την πολιτισμό, για τα προγράμματα αυτά τα οποία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα επιτυχή και έχουν αποφέρει πολλούς καρπούς, μια πραγματική προστιθέμενη αξία. Νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί ότι στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ζητήματα αυτά. Και αυτό ασφαλώς θα βοηθήσει και την Ευρώπη προκειμένου να εξέλθει της κρίσης. Πέρα από τις ευχαριστίες αυτές, θα ήθελα να πω αναφορικά με το πρόγραμμα για τον αθλητισμό. αυτό το πρόγραμμα για τον αθλητισμό και το Εράσμους ε, ακούγονται πάρα πολύ θετικά και θα ήταν πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά και την αξιοπιστία μας. Να έχουμε ένα σωστό προϋπολογισμό για προγράμματα αθλητισμού τέτοιου είδους, όπως είπε και η συνάδελφος υπάρχουν και οι συνέπειες στην υγεία, τις οποίες επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε. Όλα αυτά δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ καλή παρουσίαση, για τους καλούς στόχους, τους υποστηρίζουμε και η Επιτροπή αυτή θα ήθελε να υποστηρίξει την εργασία σας και το έργο σας. Ο Η κυρία Κώστα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πρέπει να είμαστε σύντομοι σίγουρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, το νέο πλαίσιο, στα πλαίσια του οποίου η κυρία Βασιλείου θα πρέπει να προτείνει κάποια προγράμματα προκειμένου μέσα στις τρεις αυτές κατηγορίες να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε και στη συνέχεια τίθεται και το ζήτημα της ουσίας των προτεραιοτήτων στις οποίες αναφερθήκατε αναφερόμενοι σε στόχους συγκεκριμένες δηλαδή πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, σε μια μορφή. Ως προς τη μορφή λοιπόν καταρχάς, ως προς το πλαίσιο, θα ήθελα καταρχάς να καταλάβω τα πράγματα κάπως καλύτερα. το να δημιουργήσουμε ένα πιο σαφές και οριστικό αναγνωρίσιμο πλαίσιο είναι όντως πολύ θετικό αρκεί να έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε ότι τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα. Υπάρχει η εξειδίκευση αυτή στα μέσα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε τους στόχους αλλάζοντας το πλαίσιο αυτό. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν θετικό βέβαια. Φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρόθεσή σας να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο προκειμένου να καταφέρουμε να συλλέξουμε περισσότερα χρήματα, είτε πρόκειται για τον πολιτισμό, είτε πρόκειται για την εκπαίδευση, την κατάρτιση. Πιστεύω ότι τα προγράμματά μας θα πρέπει να είναι σαφώς εστιασμένα και ξεκάθαρα. Αναφερθήκατε στην ε, EIB. Σαφώς πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης, θα πρέπει όμως πραγματικά τα επιπλέον αυτά χρήματα να βοηθούν τους ανθρώπους να έχουν αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο, να μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές, όσο και τις ίδιες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Σαφώς μπορούμε να πάμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Τώρα, για ποιο λόγο να μην δημιουργήσουμε μία καλύτερη ομαδοποίηση σε εγκάρσιο οριζόντιο επίπεδο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερο τα θετικά που έχουν διάφορα Ινστιτούτα, διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αποφεύγουμε επίσης κατά αυτόν τον τρόπο το κατακαιρματισμό. Επίσης, είπατε ότι μπορεί να κάνουμε και μία χαρτογράφηση των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. φερθεί εκτεταμένα στην κινητικότητα. Υπάρχουμε, υπάρχει όμως και η διαδικασία της ε, Μπολόνια, η οποία αυτή τη στιγμή κάπως έχει, α, ε, δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε στο παρελθόν. Στο Γιάννοφ και Τσβέα, αλλά σύντομα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς την Επιτροπό. Μία ερώτηση μάλιστα για το νέο χρηματοοικονομικό μέσο για τα προϊόντα πολιτισμού, κάτι στο οποίο αναφερθήκατε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα ειδικό οικονομικό μέσο για τέτοια προϊόντα πολιτισμού. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω αυτά που είπατε. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριο Στσβέ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθατε στην Επιτροπή μας κυρία Επίτροπε, ιδιαίτερα σήμερα. που έχετε να μας παρουσιάσετε κάποια καινούργια στοιχεία για τον τομέα της αρμοδιότητάς μας. Το τρέχον έτος είναι γενικά αρκετά ενδιαφέρον και θα καταστεί καθοριστικό για τις επόμενες ε, δημοσιονομικές προπτικές και σε άλλους ε, τομείς της πολιτικής θα καθοριστεί η πορεία μας ε, το τρέχον έτος. Αυτά που από κοινού κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το έτος θα μας συνοδεύσουν μέχρι το 2020 και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε κυρία Επιτροπέ και θέλω να σας ε, επιστήσω την προσοχή στο εξής. Καταρχάς να μην μειωθούν ε, τα χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά να αναζητηθούν ε, νέα ε, μέσα για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για τις ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επιθυμούμε πιο υψηλό προϋπολογισμό, αλλά η Επιτροπή στα τέλη του μήνα θα παρουσιάσει και τη δική της θεώρηση της κατάστασης. Θα χρειαζόμαστε και πιο πολλά για τα προγράμματα εκπαίδευσης. Εγώ είμαι υπέρ της αποδοτικότητας, προκειμένου με πιο πολλά χρήματα να πετυχαίνουμε πιο πολλά. Αλλά θα ήθελα μέχρι το 2020 όλοι να έχουν την ευκαιρία να μπορέσουν να μεταβούν στο εξωτερικό. Τέτοια κινητικότητα θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε, γιατί στην περίπτωση αυτή θα χρειαζόμαστε όχι 50% παραπάνω από όρους, 500% παραπάνω. Δεν είναι η κινητικότητα το πρόβλημα, αλλά η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτή είναι η απάντηση στην κρίση και στο ερώτημα του κατά πόσον θα είμαστε ακόμα ανταγωνιστικοί έναντι των ΗΠΑ το 2020. Εκτός μικροφώνου, η Πρόεδρος. Και έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις, επιτρέψτε μου. Είμαι υπέρ της εξοικονόμησης χρημάτων στην δίκηση, γιατί το χρήμα που, τα τις δαπάνες που δαπανούμε ε, για τη δίκηση δεν μπορούμε να, τα, να το δαπανίσουμε και στην πράξη. Πώς θέλετε λοιπόν να το κάνετε αυτό, πώς θέλετε να τα πετύχετε αυτό. Δεν θα καταργήσετε ούτε μία υπηρεσία, ούτε μία εξωτερική υπηρεσία, γιατί αυτές οι υπηρεσίες είναι που απορροφούν τα διοικητικά αυτά, τις διοικητικές αυτές δαπάνες και μάλιστα σοριδών. Πριν από κάποιες εβδομάδες είχαμε μία εκδήλωση φανταστική που μας παρουσίασε τις εξωτερικές υπηρεσίες. Πόσο μας κόστησε αυτή η εκδήλωση σε εμά που παραγγέλνουμε, που πληρώνουμε αυτές τις εξωτερικές υπηρεσίες, τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μόνο αυτά τα χρήματα σε κάποια σχολεία, για παράδειγμα. Άρα, πού θέλετε να εξοικονομήσετε τέτοιες διοικητικές δαπάνες. Αυτό το πρώτο. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην Επιτροπή ΣΟΥΡ, όπου αναφέρεται με σαφήνεια ρητά ότι τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα θα πρέπει να διατηρηθούν αυτούσια. Τρίτον, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη πολύ δύσκολο η μη επίσημη εκπαίδευση να βρει μια θέση σε αυτό το κοινό project. Πολλά προγράμματα, πολλά προβλήματα θα έχουμε αν συμφωνήσουμε να το ξεπουλήσουμε αυτό. Είμαι διατεθειμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ό,τι δεν είναι δυνατόν για να έχουμε πιο πολλά χρήματα. Αλλά αν στο τέλος καταλήξουμε να μην ξέρουμε τι πάει πού, γιατί όλα θα μπαίνουν σε ένα μεγάλο καζάνι, λυπάμαι, δεν θα έχω εμπιστοσύνη. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβεί. Θα ήθελα να ξέρω πόσα χρήματα πάνε πού, τι προβλέπετε για πού. Ποτέ, ποτέ δεν κατάλαβα ότι το πρόγραμμα για τη διαβίου μάθηση το οποίο το ε, εισάγαμε πριν από λίγο καιρό και ήμουν εισηγήτρια, τώρα ξαφνικά. Γιατί πρόκειται για πρόγραμμα ομπρέλα. Τώρα, είτε ονομάζεται μάθηση, είτε ονομάζεται ε, εκπαίδευση νεολαία, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι το κατά πόσον μπορεί να υπάρχουν καλύτερε συνδέσεις στο εσωτερικό του προγράμματος, αν υπάρχει οριζόντια συνεργασία. Αυτό μπορεί να γίνει και με το παλαιό πρόγραμμα όμως, αν υπάρχει θέληση. Γι' αυτό Ευχαριστώ να σας πιστέψω, να πιστέψω και τους υπαλλήλους σας ότι όλα αυτά θα καταστούν δυνατά με το νέο πρόγραμμα, αλλά δεν έχω πιστεί ακόμα. Θα ήθελα να σας επενέσω όμως για την συμπερίληψη της διαβίου μάθησης σε ό,τι αφορά τα master, τα προγράμματα masters. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν μπορούμε να τα πετύχουμε εμείς Την προηγούμενη φορά συζητήσαμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε τα σχετικά μέσα. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός ο τρόπος για το EIB που επιλέξατε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, αλλά και το Εράσμος Μούντους θα μπορούσε να ενταχθεί στη διαβίου μάθηση. Γιατί... Αυτά, αυτά ήθελα να σας αναφέρω ως παρατηρήσεις. Συμφωνώ με αυτά που ακούστηκαν και θα ήθελα να μας διευκρινίσετε λίγο αυτά που σας ρωτήσαμε. Έχετε το λόγο, κυρία Επιτροπέ. Uh, θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω κάτι γιατί ίσως υπήρξε μια παρανόηση. Ξέρετε ότι μερικές φορές έχουμε μια παγιωμένη αντίληψη στο μυαλό μας και δεν ακούμε τους άλλους προσεκτικά. Ουδέποτε είπα ότι θα συνδυάσω σε ένα πρόγραμμα τον πολιτισμό και τα μίντια το πρόγραμμα Media και το πρόγραμμα για, την, για τον πολιτισμό. Κάποιος το είπε αυτό βέβαια εδώ πέρα. Θα έχουμε ένα πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης θα έχουν κοινό προπολογισμό, κοινή διαχείριση. Θα εξακολουθούν να είναι δύο ξεχωριστά προγράμματα. Και είπα ότι αν καταφέρω να εξασφαλίσω περισσότερα χρήματα, τότε θα υπάρχει και ο άλλος τομέας για τον πολιτισμό και τις δημιουργικές επιχειρήσεις. Και στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει ένα ταμείο εγγύησεων προκειμένου να δίνονται στις επιχειρήσεις αυτές κάποια δάνεια γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα για τις επιχειρήσεις αυτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας να έχουν πρόσβαση σε δανειοδότηση. Επίσης, έχω την εντύπωση, δεν μπορώ να είμαι απόλυτα πεπισμένη βέβαια, αλλά μερικές φορές η γλώσσα του σώματος μιλάει από μόνη της. Και το λέω αυτό γιατί όταν μιλούσα με τους συνομιλητές μου από το τομέα του προπολογισμού έβλεπα ότι για τον αθλητισμό ήταν λίγο διστακτική για ποιο λόγο να αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο, μπορεί να ενταχθεί στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση. Σιγά σιγά όμως είδα ότι κάπως χαλάρωναν και ότι άλλαζαν στάση. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι κατάφερα να τους πείσω, είμαι όμως περισσότερο αισιόδοξη τώρα από ότι ήμουν πριν από ένα μήνα. Α το αποδεχτούμε λοιπόν αυτό και προφανώ εσείς θα πρέπει να εφηραματίσετε το δικό σα το ρόλο. Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση. Όπως σα είπα, ο στόχος μου για την εκπαίδευση, την νεολαία και την κατάρτιση δεν είναι να έχουμε τις ίδιες δράσεις με τα ίδια χρήματα. Στόχος μου είναι η απλούστευση και ο περιορισμός του διοικητικού άχθους προκειμένου να καταφέρω να τους δείξω ότι όντως εμείς από τη δική μας πλευρά κάνουμε μια σημαντική προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουν να μας δώσουν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την νεολαία. Και για αυτό το ζήτημα είμαι αισιόδοξη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε. Ακούστηκε και μια άλλη παρατήρηση, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να καλύψουμε το, την ενδιάμεση αυτή κατηγορία των ανθρώπων που βρίσκονται μεταξύ του σχολείου και του πανεπιστημίου. Η κυρία Μακλάρε νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό. Σίγουρα επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αποκριθεί στο αίτημα αυτό και θα πρέπει από την άλλη όμως να έχουμε και κάποια προγράμματα κινητικότητας προκειμένου οι άνθρωποι αφού να μπορούν να βρουν κάποια εργασία τουλάχιστον ένα πρόγραμμα κατάρτιση σε μια επιχείρηση. Και δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που είπαμε και πριν από λίγο, να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε, πώς μπορούμε μάλλον να καλύψουμε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα πανεπιστήμια και την αγορά εργασίας. Εκεί έγκυται το πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε πάρα πολλούς πτυχιούχους οι οποίοι είναι άνεργοι πρόθεσή μας δεν είναι να υποκαταστήσουμε αυτό το οποίο θέλουν αυτοί να σπουδάσουν με αυτό που θα θέλαμε εμείς να σπουδάσουν. Στόχος μας είναι να τους προσφέρουμε μια καλύτερη ενημέρωση. Όταν δηλαδή ξεκινάνε τι σπουδέ τους θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ενημέρωση που θα τους επιτρέψει να κάνουν μια σωστή επιλογή του τι πιστεύουν ότι θέλουν να σπουδάσουν. Και βέβαια αφού ολοκληρώσουν τις σπουδέ τους θα πρέπει να συμπληρώσουμε τις σπουδέ τους με μια εμπειρία και με κάποιες εγκάρσεις δεξιότητες, οι οποίες όπως σας είπα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και έρχομαι τώρα στο ερώτημα της κυρίας Παλιαδέλη. Κατ' εμένα είναι πολύ βασικό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις ανθρωπιστικές σπουδές διότι με το να σπουδάσουν ανθρωπιστικές σπουδές δεν θα μπορέσουν να εργοδοτηθούν. Το θέμα είναι ότι οι ανθρωπιστικέ σπουδέ που παρακολουθούν τα παιδιά μα πρέπει να είναι η βάση τους και πέραν από αυτόν πρέπει να τους δώσουμε τι ευκαιρίε να συμπληρώσουν αυτά τα οποία έμαθα στο πανεπιστήμιο με όλα τα άλλα τα οποία θα χρειαστούν. Και αυτό θα το επιτύχουμε με, τα, ε, με apprentices, ε, με, training abroad, με, ε, το mobility, language learning, όλα αυτά τα οποία είχαμε πει. Και πρέπει να σας να πω ότι τα προγράμματα μας για τους ερευνητές, όπως είναι το Marie Curie, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα, δεν περιορίζεται στις θετικές επιστήμες. Είναι μια λανθασμένη εντύπωση. Απλούστατα, ίσως ξεκινώντας από αυτήν την λαθασμένη εντύπωση, δεν έχουμε πολλές αιτήσει για αυτόν το, αυτόν το πεδίο της έρευνας. Αλλά είναι ανοιχτό το Marie Curie είναι ανοιχτό για όλους τους τύπους έρευνας. Γι' αυτό θα πρέπει κάπως να το, ε, να το κάνουμε πιο γνωστό ε, σε όλους οι οποίοι ενδιαφέρονται για έρευνα. Είναι θέμα νομίζω το πώς διαφωτίζουμε τον κόσμο για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Ε, για τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων είναι μια δύσκολη, είναι μια δύσκολη εργασία για την οποία πρέπει να υπάρξει απόλυτη συνεργασία μεταξύ των χωρών των κρατών μελών ε, και, των Βρυξελών. Διότι αποφασίζουμε για ορισμένες βασικές πολιτικές. Αυτές οι βασικές πολιτικές θα πρέπει να εφαρμοστούν και ίσως με τις τροποποιήσεις που χρειάζονται για, να, για την ε, ε, συγκεκριμένη περίπτωση αλλά δεν μπορεί η κάθε χώρα να, να, βάζει δικές της πολιτικές όσον αφορά την ανώτερη εκπαίδευση. Πρέπει όλοι μας να ακολουθήσουμε τις βασικές πολιτικές τις οποίες έχουμε αποφασίσει ή θα αποφασίσουμε. Διότι όπως σας είπα ε, θα έχουμε τη νέα μας πρωτοβουλία για τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων τον Οκτώβριο και ελπίζω αυτό να αποτελέσει ε, έναν πολύ καλό θέμα για συζήτηση διότι είναι πολύ βασικό για όλες τις χώρες. Διότι πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο λειτουργεί σε αυτές τις χώρες και είναι επιτυχημένες και τι είναι αυτό που δεν λειτουργεί και να μάθουμε η μία από την άλλη ε, συγκρίνοντας τα συστήματά μας. Ε, the question of has been raised in relation... Το ζήτημα του φόρου προστιθέμενης αξίας έχει τεθεί σε σχέση με τον αθλητισμό. Ο φόρος προστιθέμενη αξία αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, όπω το ξέρετε. Δεν μπορούμε εμείς από εδώ, από τις Βρυξέλλε, να πούμε στα κράτη-μέλη τι θα κάνουν με τον ΦΠΑ. Και για παράδειγμα, ξέρω ότι το ζήτημα αυτό ετέθη ιδιαίτερα έντονα σε σχέση με τα βιβλία, τα έντυπα βιβλία, σε σχέση με τα ηλεκτρονικά βιβλία και έχει ξεκινήσει ένα κίνημα από τη Γαλλία κυρίως, προκειμένου ο μειωμένος ΦΠΑ που ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένα κράτη-μέλη για τα έντυπα βιβλία στα ηλεκτρονικά βιβλία, τα βιβλία στο διαδίκτυο. Πρέπει να σας πω όμως ότι στην Επιτροπή, που στην Επιτροπή που συζητήσαμε το ζήτημα αυτό μόνο η Γαλλία υποστήριξε αυτή την ιδέα. Για να αλλάξουν οι κανόνες χρειάζεται ομοφωνία. Για να αλλάξουν οι κανόνες του φόρου προσθέμενης αξίας απαιτείται ομοφωνία. Και βέβαια το εγχείρημα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και σαφώς το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε εξαίρεση δίνεται από οποιοδήποτε κράτος μέλος για οποιαδήποτε αθλητική οργάνωση ομοσπονδία. Ε, Σαφώ και εγώ θα ήλπιζα να μπορούσε να ίσχυε αυτό σε όλε τι χώρε, αλλά δυστυχώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, τουλάχιστον τώρα. Και να πω κάτι ακόμα. Αναφέρθηκα σε συνέργειε. Όταν αναφέρομαι σε συνέργειε, αναφέρομαι και σε συνέργειε ανάμεσα στα προγράμματα διαβίου μάθησης, ανάμεσα στο κοινωνικό ταμείο και με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ξέρετε ότι και τα δύο αυτά διαφορετικά ταμεία τα πανούνε πολλά χρήματα και νομίζω ότι είμαστε ο μόνος τομέας, δηλαδή η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, όπου υπάρχει μία επαρκή ζήτηση για όλα αυτά τα χρήματα, για όλους αυτούς τους πόρους και τα κονδύλια. Δυστυχώς όμως στο παρελθόν ουδέποτε υπήρξε ένα συντονισμός πολιτικών ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση περιφερειακής ανάπτυξης, απασχόλησης και εκπαίδευσης. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει μία επιτροπή η οποία θα αποφασίζει πώς θα συντονίζουμε αυτούς τους τρεις τομείς πολιτικής προκειμένου όλοι να στοχεύουμε προς τις ίδιες πολιτικές. Αν στόχος μας είναι να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα πρέπει να καταφέρουμε να συγκεράσουμε τις προσπάθειές μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι απάντησα σε ερωτήσεις. Υπάρχει το δικό μου το ερώτημα, λέει η κυρία Πάκ, για τη διοίκηση. Μα νομίζω ότι αναφέρθηκα σε αυτό. Αν τα κράτη-μέλη ζητούν να μειωθούν οι διοικητικές δαπάνε να μειωθούν όλες οι υποστηρικτικές διοικητικές δραστηριότητες, να γίνουν τα πράγματα πιο διαφανή και πιο απλά. Προφανώς δεν μπορώ εγώ να παραβλέψω τα αιτήματα αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να βασίζομαι και στα κράτη-μέλη προκειμένου να έχω περισσότερους πόρους. Οπότε πρέπει να τους δείξω ότι όντως ανταποκρίνομαι στα αιτήματά τους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα στη δική σας, στη Γερμανία ή στην Ιταλία, υπάρχουν τρεις διαφορετικές υπηρεσίες τις οποίες εμείς χρηματοδοτούμε και η μία δεν ξέρει τι δουλειά κάνει η άλλη. Πήγα στη Φλωρεντία και είχαμε διοργανώσει εκεί πέρα μια σημαντική συνδιάσκεψη. Άκουσα ένα πρώτο λόγο και θεώρησα ότι ο πρώτος αυτός λόγος κάλυπτε όλες τις υπηρεσίες που είχε η χώρα αυτή αλλά μου είπαν ότι όχι, πρέπει να ακούσουμε και την άλλη υπηρεσία, τον άλλον οργανισμό, γιατί έχουν αυτοί, είχαν και αυτοί να πούνε κάτι παραπάνω. Οι χώρες αυτές που έχουν πάνω από έναν οργανισμό, πάνω από μία υπηρεσία, θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να καταφέρουν να γίνουν λίγο πιο αποτελεσματικοί, να καταφέρουν να έχουν ε, ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και ορατότητας. Καταλαβαίνετε ότι θα καταφέρουμε να, γίνουμε, να προβληθούμε πολύ περισσότερο αν πετύχουμε αυτές τις συνέργειες. Πώς είπατε? Για την ανεπίσημη μη επίσημη κατάρτιση. Ναι, αυτό αποτελεί προτεραιότητα για μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να σαρίσουμε από τους ε, νέους, από τους εθελοντές, τα προγράμματα γεννητικότητας σε ό,τι αφορά την επίσημη και τη μη επίσημη ε, εκπαίδευση και κατάρτιση και για να το αποδείξουμε αυτό θα εγκρίνουμε μια σύσταση σύντομα για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις μορφές εκπαίδευσης και επίσης ε, να διαβρύνουμε το Europass, το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο, όχι μόνο να περιλαμβάνει τις ακαδημικές ε, ικανότητες, αλλά και τη μη τυπική και ατυπική μορφή εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχουμε ακόμα και μετά θα δώσω το λόγο πάλι στον Μπόης. Κυρία Μποσκούρτ. Όχι δεν απαντήθηκε το ερώτημά μου για τα παράνομα στοιχήματα και για τα πρακτορία. Mark, uh, Mrs. και τους μάνατζερ των παικτών. Ε, αναφέρθηκα στο ανοιχτό ταμείο για το ποδόσφαιρο που δραστηριοποιείται στην Βοσνία Ερσεγοβίνη. All the, all the όλες τις δράσεις που αναφέρατε, για παράδειγμα, παράνομος στοιχηματισμός, ε, μάνατζερ επεκτών, είναι προβλήματα σοβαρότατα και πολύ σχηδή. Και δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι με τη διοργάνωση ενός συνεδρίου θα λύσουμε το πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση. Τουλάχιστον θα μάθουμε περισσότερα πράγματα και για το πρόβλημα και για τις ιδιαιτερότητές του. Και για να το καταφέρουμε αυτό φυσικά και πρέπει να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, με την ΟΕΦΑ. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Διότι ο καθένας μας έχει ένα κομμάτι της ε, πληροφορίας. Πρέπει να ενώσουμε τα κομμάτια για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θα το λύσουμε ούτε σε ένα χρόνο ούτε με ένα συνέδριο. Θα χρειαστεί χρόνος. Παράνομος στοιχηματισμό. Για παράδειγμα είναι κάτι που έχει απασχολήσει τον Επίτροπο Μπαρνιέ που ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για τον ε, online στοιχηματισμό και η κυρία Μάλστρομ έχει αναλάβει επίσης μια πρωτοβουλία για την ε, διαφθορά εν γέννη αλλά εγώ κατάφερα να συμπεριλάβει η κυρία Μάλστρομ στην πρωτοβουλία της τον αθλητισμό τη διαφθορά στον αθλητισμό. Όπως βλέπετε λοιπόν, αν αυτό το πρόβλημα που έχουμε στον αθλητισμό το επεκτείνουμε και στις άλλες ε, γενικές διευθύνσεις που έχουν κάποιους παρόμοιους τομείς αρμοδιότητας, μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα. Οι πρωτοβουλίες που αναφέρατε για την υγεία και τον αθλητισμό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εξού και οι υπηρεσίες μου άρχισαν επί παραδείγματα να συνεργάζονται με τις υπηρεσίε του Επιτρόπου Ντάλι για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα τον αθλητισμό για την υγεία στα σχολεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε εταιρικέ σχέσεις ακόμη και μέσα στην ίδια την Κομισιόν. Γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα της μίας επιτροπής για να συμπληρώσουμε τα μέσα της άλλης επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για τον προϋπολογισμό αν ενώσουμε αυτό που έχει εκείνος με αυτό που έχω εγώ, μπορεί να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Shortly, Triple, shortly, shortly, Πάρα πολύ σύντομη κυρία Τρίπελ και μετά ο κύριος Μπόρης. Να προσθέσω κάτι για την αναδιάρθρωση των οργανισμών, πολιτικό σχόλιο. Ε, αναδιάρθρωση των οργανισμών σε επίπεδο κρατών μελών. Αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μείωση του διοικητικού άχθους και μεγαλύτερη διαφάνεια, αυτό για μένα είναι καλό. Αλλά για πολιτικούς λόγους νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι λίγο πολύ είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και του Συμβουλίου. Δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί εμάς μας ζητούν να κάνουμε περικοπές. Αλλά αυτή είναι υπεύθυνη και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κύριος Μπόρις τώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι αυτά που μας είπε μόλις η Ευρωπαϊκή η Επιτροπός για τις ε, προτεραιότητες και την στρατηγική μας θα πρέπει να ε, κερδιθεί με αγώνα, με θετική άποψη. Θεωρώ ότι ο ορισμός των μέσων για τον αθλητισμό και την εκπαίδευση. και να σας πω, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και σε ό,τι αφορά το lifelong learning, το media και όλα αυτά, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την περιφερειακή ανάπτυξη, όπου δεν έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια, έχουμε δισεκατομμύρια ευρώ για διάφορα μέτρα Δεν ξέρω αν ε, είναι στο χέρι σας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία γιατί από την δική σας ε, ε, ικανότητα θα εξαρτηθεί το μέλλον αυτών των πολιτικών. Αν το... όλα αυτά τα προγράμματα θα στεφθούν με επιτυχία. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Μία μικρή σύσταση. Μιλήσατε για την διαφθορά στον αθλητισμό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι με το πρόβλημα αυτό, το οποίο έχει πολλές διαφορετικές όψεις και σε διάφορα επίπεδα, θα πρέπει ίσως να ψηφιστεί στην Επιτροπή Γιούρη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις στον τομέα του αθλητισμού. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτό προκειμένου να υπάρχει ε, ε, εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επίτροπος να απαντήσω στην παρατήρησή σας. Μα ακριβώ γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με την Επίτροπο Μάλστρομ. Προφανώς εμένα με ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό, αλλά αυτή ουσιαστικά γνωρίζει ποιες είναι νομικές δυνατότητες για να γίνει κάτι στην πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε λοιπόν και με εσά, αλλά και με άλλες επιτροπές προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Μια τελευταία παρατηρήση. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνετε. Αν δούμε την έκθεση της Επιτροπής ΣΟΥΡ, βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες. Και το λέω αυτό γιατί στην έκθεση ΣΟΥΡ υπογραμμίστηκε πάρα πολύ έντονα το ζήτημα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης του πολιτισμού, του αθλητισμού. Για τον αθλητισμό ήλπιζα ότι θα είχε γίνει μια πιο ισχυρή δήλωση, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να σκεφτεί κανείς. Πιστεύω πάντως ότι στον τομέα μας θα καταφέρουμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα, σαφώς θα πρέπει να δώσουμε αγώνα. Ξέρω ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη κάνουν περικοπές στον προπολογισμό τους. Για παράδειγμα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγα στις κάτω χώρες και γινόταν εκεί πέρα μια πολύ μεγάλη διαδήλωση κατά των περικοπών στον τομέα του πολιτισμού και ανάλογες έχουν συμβεί σε πολλά κράτη-μέλη. Γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι σαφώς οι διαπραγματεύσεις θα είναι πολύ σκληρές με το Συμβούλιο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και γι' αυτό όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτά αποτελέσματα. Γιατί ξέρω ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε ουσιαστικά τους ίδιους στόχους και θέλουμε να πετύχουμε από κοινού τους στόχους αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Μια τελευταία παρατήρηση. Η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών αυτών τομέων ως προς τον υπολογισμό καταλαβαίνετε ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά, πρέπει εμείς να μειώσουμε τον προπολογισμό μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι ο συντονισμός είναι η μαγική λύση και να βρισκόμαστε μετά με λιγότερα χρήματα όμως. Σας ευχαριστούμε πολύ και προσβλέπουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τη δικό σας το έγγραφο στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Okay. Colleagues, you can, you can stay, yeah? Μα αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να μείνετε, ξέρετε. Ο κύριος Λόχεργκάρτ είναι ο συγγητής για το επόμενο ζήτημα, προπολογισμός 2012. Πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Ξέρετε ότι η τοποθέτηση του Συμβουλίου προβλέπεται για τις 25, για τις 29 μάλλον Ιουλίου. Νομίζω ότι περισσότεροι θα είμαστε ήδη τότε σε διακοπές και γι' αυτό το λόγο οι συντονιστές αποφάσισαν ότι η Επιτροπή Πολιτισμού, ακούστε με παρακαλώ, είναι σημαντικό. Δεν είμαστε στο σχολείο εδώ πέρα, με να συμπεριφέρομαι έτσι. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα ψηφίσει τις τροπολογίες για τον προπολογισμό στις 14 Ιουλίου. Προτού λάβουμε δηλαδή τη δήλωση Συμβουλίου, θα ψηφίσουμε για την πρόταση της Επιτροπής που έχει τροποποιήσει ο κύριος Λόχεγκάρντ. Οι τροπολογίες θα υποβληθούν και θα ψηφιστούν στα αγγλικά για τεχνικούς λόγους. Δεν μπορούμε να έχουμε τη μετάφραση νωρίτερα. Και ο κύριος Μόρτεν Λόκεγκάρτ θα υποβάλει, θα παρουσιάσει στις 14 Ιουλίου όλες τις τροπολογίες που θα έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή μας και θα είμαστε στη συνέχεια σε θέση να ανακτήσουμε κάπως τον προπολογισμό και τους τομείς εκείνους που το Συμβούλιο θέλει μείωση. Αν είστε ικανοποιημένοι λοιπόν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλετε να ανακτήσετε τον προπολογισμό σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίσει να μειώσει τον προπολογισμό, δεν χρειάζεται εσείς να υποβάλλετε ξεχωριστές τροπολογίες και θα το κάνει για σας ο κύριος Λόκεγκάρτ. Αν θέλετε τώρα να αλλάξετε το σχέδιο προπολογισμού της Επιτροπής, θα πρέπει να υποβάλλετε στα αγγλικά τις τροπολογίες σας μέσα 27 Ιουνίου. 27 Ιουνίου, μην το ξεχνάτε αυτό. Κύριε Λόκεγκαρτ, έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που τονίσατε ότι είναι σημαντική η δουλειά μου. Έτσι θα τη σκεδάσουμε ακόμη περισσότερο. Και όπως ε, είπε η Πρόεδρος, ε, εσείς μπορείτε να πάτε διακοπές και εγώ θα δουλεύω. Τι να κάνουμε. Τα επόμενα λεπτά πάντως ε, μπορείτε να μου αφιερώσετε λίγο την προσοχή σας. Ε, ήδη δύο φορές σε προηγούμενες συναντήσεις μας έχουμε πει ότι καταφέραμε να βάλουμε το δικό μας αποτύπωμα και στην τελική περσινή συμφωνία με τα 18 εκατομμύρια παραπάνω για την ε, ηλεκτρονική μάθηση και τα 3 έξτρα εκατομμύρια ευρώ για τον αθλητισμό. Καλές εξελίξεις αυτές, αλλά βέβαια μπορούμε να τα καταφέρουμε φέτος ακόμη καλύτερα ιδίως αν επικεντρώσουμε τις προτεραιότητές μας ε, καλύτερα σε σχέση με πέρυσι και αυτή είναι και η βασική μου παρατήρηση. Νομίζω ότι υπήρξαμε αλλά μπορούμε να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι ακούγοντας μάλιστα την Επιτρόπο και αν έχουμε την στήριξή της ε, θα τα καταφέρουμε πιστεύω. Έχουμε δυνατότητες, αλλά επαναλαμβάνω πρέπει να είναι σαφείς οι στόχοι μας και βέβαια θα πρέπει να σεβαστούμε του περιορισμένου πόρου που υπάρχουν, τα επιπλέον κονδύλια που είναι μέσα στα περιθώρια για φέτο. Αναφέρθηκα ε, σε αυτά την τελευταία φορά. Είναι 150 εκατομμύρια ε, για την κατηγορία 1α και 15 για την κατηγορία 3β. Ε, δεν ξέρω αν θα τα πάρουμε όλα αυτά τα χρήματα, αλλά αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, για τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οι προτεραιότητες μας λοιπόν πρέπει να εστιαστούν σε δύο θέματα κυρίως. Πρώτα απ' όλα η διαβίου μάθηση και βέβαια ο αθλητισμός. Με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία που είχαμε και στις συνομιλίες που έχουμε κάνει, νομίζω, τουλάχιστον εγώ αυτό διαστάθηκα ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση. Περιμένουμε τη συνένεση αυτή να συνεχίζει, να υπάρχει. Ελπίζουμε τουλάχιστον. Συγκεκριμένε τώρα τροπολογίες, αν τις δείτε, θα δείτε ότι έχω κάνει και για τις δύο κατηγορίες και για την προπαρασκευαστική ενέργεια για τον αθλητισμό και για τη διαβίου μάθηση. Δεν μπορείτε να, να μην τις θεωρήσετε οριστικές αυτές τις τροπολογίες, απλά θέλω να δείτε περίπου τη λογική που ακολουθώ. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, αλλά ουσιαστικά οι πρώτες ιδέες μου είναι αυτές. Σε σχέση με τα επίπεδα, αν δείτε Λοιπόν, θα δείτε ότι προτείνω 45 εκατομμύρια παραπάνω για τις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων για τη διαβίου μάθηση. και θα γίνει με τις πληρωμές θα πείτε κάποιοι, γιατί δεν έχουμε στοιχεία εκεί. Απλά ζητήσαμε να μας πει η Επιτροπή και μας είπε ότι 30 εκατομμύρια περίπου μπορεί για το πρώτο έτος να δαπανίσει. Άρα Το επίπεδο είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια. Αν έχουμε μία ανάλυση πόρων για 45 εκατομμύρια. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι μία πρόταση διαπραγμάτευση. Θα πρέπει πάντως να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα σε σχέση με τη διαβίου και με τους στόχους μας. Νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες να πετύχουμε πολλά. Βέβαια, για το τελικό νούμερο θα τα ξαναπούμε, αλλά πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Δεύτερο τώρα, προπαρασκευαστική ενέργεια για το πρόγραμμα για τον αθλητισμό. Και εδώ πρόκειται απλά για υπόδειξη. Έχω βάλει το νούμερο 6 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσά θα θέλουν ε, ένα μεγαλύτερο νούμερο. Μπορούμε να το συζητήσουμε βέβαια αυτό, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι που μπορούμε να συμφωνήσουμε, εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Να έχουμε μία τροπολογία θα έλεγα Έχω μιλήσει με μερικούς από εσά και νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να αναμένουμε μια καλή συνένεση. Δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, οπότε δεν έχω κάνει προτάσεις συγκεκριμένες, αλλά θα προσπαθήσω να προσθέσω δικά σας πιλωτικά προγράμματα ή προπαρασκευαστικές ενέργειες σε αυτήν την προπαρασκευαστική ενέργεια. Ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Επίσης, έχω προσθέσει δύο πράγματα, πιλωτικά προγράμματα για εταιρικές σχέσεις γνώσης. Βλέπετε ότι μιλάμε αύξηση των υφιστάμενων πιλωτικών προγραμμάτων που την χάνουν μεγάλης υποστήριξη από την Κομισιόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζει πάρα πολύ την ε, στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Οι εταιρικέ σχέσει γνώση αναφέρεται αυτό ε, στην ε, συγκεκριμένη στρατηγική. Θέλουμε να βελτιώσουμε την έρευνα, την καινοτομία, να έχουμε ένα εξεχρονισμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Όλοι συμφωνούμε. Άρα πρέπει να μπουν και κάποια έστω και μικρά ποσά και στον προπολογισμό τη επόμενη χρονιά. Γι' αυτό και προτείνω τη σχετική τροπολογία. Τέλο, τέταρτη τροπολογία. Ενημέρωση για τα ΜΜΕ είναι η γραμμή. Νομίζω το είχα ξαναπεί. Μιλάμε για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια δημοσιογράφου. Αυτά εμπίπτουν σε, αυτή την, ε, σε αυτό το κονδύλιο του προπολογισμού. Για να πω δύο λόγια πάνω σε αυτό Στόχος είναι να ενημερωθούν οι δημοσιογράφοι για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τέτοια σεμινάρια αποδείχθηκαν ότι είναι πολύ δημοφιλή. Πάντοτε υπήρχαν υπεράριθμες κρατήσεις και βλέπουμε ότι το επίπεδο των γνώσεων των δημοσιογράφων είναι ένα τομέα πολύ συγκεκριμένο πάνω στον οποίο πρέπει να καταβάλουμε με μεγαλύτερε προσπάθειε να βοηθήσουμε του δημοσιογράφου να κατανοήσουν το πολύπλοκο αυτό σύστημα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα στον τομέα αυτό και να είμαστε και πιο φιλόδοξοι. Γι' αυτό και έχω καταθέσει τη σχετική τροπολογία. Ένα τελευταίο εξίσου σημαντικό όμω ε, ζήτημα είναι, και θέλω να επιστρέψω την προσοχή τη Επιτροπή σα σε αυτό, είναι ο προπολογισμό για την επικοινωνία. Νομίζω ότι πράγματι πετύχαμε πολλά στον τομέα της εκπαίδευσης και συνεργασία με τη ΓΔ ΙΕΚ. Και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τα κέρδη και το ωφέλη που αποκομίσαμε κατά την περσινή χρονιά και ίσως και φέτος πετύχουμε κάποια πράγματα. Στρεφόμενος προς την ΓΔ ΚΟΜ τώρα δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο. Τίποτα δεν καταφέραμε τα τελευταία δύο χρόνια. Και βέβαια αυτό είναι ανησυχητικό. Και με απασχόλησα το γιατί. Αν δείτε λοιπόν τι περιλαμβάνει το θεματολόγιο ε, στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο μας δύο φορές και πέρσι και φέτος έχουμε εγκρίνει προγράμματα για τη διασυνοριακή δημοσιογραφία και την έρευνα και τέλος πάντων ε, βλέπουμε ότι έχει διαγραφεί αυτό το ε, project. Υπήρξε επίσης και υπάρχει ακόμη αυτή η διαδικασία ένα χρόνο τώρα, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα και το Κοινοβούλιο έχει παραπονεθεί στην Επιτροπή Παραπολογισμών για αυτό το θέμα, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποδώσει αυτή η προσπάθεια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει με αυτό το project και να βρούμε μια λύση. Κάποιοι θα έλεγα ηγετικέ δυνάμει έχουν υποσχεθεί ότι θα προχωρήσουμε, αλλά τέλο πάντων δεν έχουμε ακόμη κάποιο απτό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι καταφέραμε να υπάρξουν κάποιες αυξήσεις ε, για τους ευρωπαϊκούς δημόσιους χώρους, 1,1 έξτρα εκατομμύριο και 1,5 εκατομμύριο έξτρα για τα κέντρα πληροφοριών. Πετύχαμε λοιπόν η ΓΑΜΑ να έχει περισσότερα κονδύλια, αλλά δεν μας έδωσαν αυτοί κάτι ως αντάλλαγμα και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ικανοποιητικό αυτό. Ίσως θυμάστε κάποιοι από εσάς, μάλιστα κάποιοι Γερμανοί συνάδελφοι στην Επιτροπή παραοικολογισμών ε, είχαν ε, ζητήσει να έχουμε ένα αποθεματικό γύρω στα Χριστούγεννα το είχαν ζητήσει αυτό για τη στρατηγική για τον τομέα αυτό των επικοινωνιών. Το Γενάρη συναντηθήκαμε με την Κομισιόν, αλλά δεν υπήρχε στρατηγική, άρα μπορεί κανείς να αναρωτηθεί γιατί ήρθε το αποθεματικό, ήρθε πάντως. Έγινε αυτό, αλλά της ουσίας μηδέν. Τέλος, στην ίδια συνάντηση του Γενάρη, η Επιτροπή μας έδωσε ότι το TVNet EU, ε, το δίκτυο αυτό, που είχε 8,5 εκατομμύρια ευρώ στον προπολισμό, έκλεισε. Έκλεισε χωρίς κανένα σχόλιο όμως και χωρίς να ζητηθεί γνώμη μας. Διερωτώ με. Τα χρήματα αυτά που πήγαν. Έχω κάποιες ιδέες, ίσως μπορούμε να τις συζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό υπηρετούνται οι στόχοι που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να ολοκληρώσω, έχω και άλλα παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να σας ε, κουράσω. Για να συνοψίσω λοιπόν. Η Επιτροπή μας νομίζω ότι αξίζει καλύτερη μεταχείριση στον τομέα αυτό. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική, πρέπει εμείς ως Κοινοβούλιο να μπορούμε να συμμετέχουμε στον τομέα αυτό. και δεν θα πρέπει να έχουμε έλλειψη συνεργασίας από πλευράς ε, κομισιών. Υπήρχε και μια συνάντηση τη θεσμική ομάδα εργασία την προηγούμενη εβδομάδα και εμεί από πλευρά Κοινοβουλίου προσπαθήσαμε να ιεραρχήσουμε κάπω τι προτεραιότητε για το 2012. Δεν πετύχαμε τίποτα όμω. Ε, δεν ξέρω αν περίμενε και κανεί ε, να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Εμεί όμω τα αιτήματά μα τα υποβάλαμε. Η Επιτροπή μας νομίζω ότι πρέπει να υψώσει το ανάστημά τη να ζητήσει, διεκδικήσει αυτά που θέλει και θα έλεγα να ε, προσπαθήσουμε σε μια συνεδρία των συντονιστών να επιλύσουμε το πρόβλημα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το φετινό προϋπολογισμό, το προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σπελέτ. Ευχαριστώ Ντόρις. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος να ανακοινώσω ότι η ομάδα μας θα ήθελε να υποστηρίξει τον εισηγητή, ιδιαίτερα στις προσπάθειες που καταβάλει για διάφορα ζητήματα συγκεκριμένα στην διαβιομάθηση, στον αθλητισμό, 100% υποστηρίξη δηλαδή, στην τακτική του. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόταση αύξηση του προπολογισμού για την διαβίου μάθηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιδείξουμε φιλόδοξη στάση. Κατά δεύτερον, αυτό που ανακοίνωσε και η Πρόεδρος, φυσικά εμπιστευόμαστε απόλυτα τις δυνάμεις σας και τις προσπάθειες που καταβάλλετε για να εξισορροπήσετε τις περικοπές του προϋπολογισμού που θα προτείνει η Επιτροπή και να επανακαταθέσετε προτάσεις της Επιτροπής μας. Μία μικρή παρατηρήση σε ό,τι αφορά την τρίτη τροπολογία για τις εταιρικές σχέσεις γνώσης. Φυσικά το υποστηρίζουμε, αλλά πρόκειται για συμβολικό ποσό. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο και καταλαβαίνω γιατί, γιατί δεν υπάρχουν φυσικά χρήματα. Αλλά να υπενθυμίσω αυτό που είπε η Επίτροπος πριν από λίγα λεπτά. Αναφέρθηκε σε συνέργειες με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να ήταν αποδοτικός ο τρόπος αυτός. προκειμένου να εξευρεθούν περαιτέρω κονδύλια για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Αυτές οι βασικές μου παρατηρήσεις. Ε, γενικά υποστηρίζουμε ε, τις ε, προσπάθειές σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Καμέβερτ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι και εγώ μπορώ το δίχω άλλο να υποστηρίξω τι προτάσεις του κ. Λόκεγκαρτ, αλλά στον αθλητισμό θα ήθελα μετά από αυτά που ζητήσαμε και το προηγούμενο έτος, που ζητήσαμε 10 εκατομμύρια, το προηγούμενο έτος ζητήσαμε 10 εκατομμύρια. Ξέρουμε ότι στι διαπραγματεύσει τα πράγματα πάντα έτσι. Ζητάμε πιο πολλά και παίρνουμε λίγα. Τελικά ε, Αν ζητήσουμε όχι 10 αλλά 6 θα μας δώσουν 1,5 εκατομμύριο. Ίσως λοιπόν να σκεφτούμε για να ακολουθήσουμε και τη γραμμή του προηγούμενου έτους, να παραμείνουμε στα ίδια επίπεδα, να ξαναζητήσουμε αυτά που ζητήσαμε την προηγούμενο έτος. Γιατί μου προκαλεί έκπληξη. Μα είπε η Επιτροπό Βασιλείου πόσο σημαντικό είναι ο κλάδο αυτό και ότι θα ήθελε να υπάρχει και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Μου προκαλεί έκπληξη που η Κομισιόν για το τρέχον έτος ε, δεν ε, έδωσε κονδύλια για το τομέα αυτό. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να μην ήταν το ποσό αυτό που θέλαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν υψηλό. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να σκεφτούμε από τακτικής ε, άποψης τι ενδείκνυται. 6 εκατομμύρια ή μήπως να ακολουθήσουμε ε, την ε, γραμμή της προηγούμενης χρονιάς και να ζητήσουμε 10. Αυτά λοιπόν από δικής μου πλευράς. Ευχαριστώ, κυρία Τρούπελ, λέει η πρόεδρο. Ευχαριστώ, Ντόρις. Ναι, εμεί ω πράσινοι υποστηρίζουμε επίσης την πρόταση του κύριου Λόκεγκάρ, του Μόρτεν, Συμφωνώ με την κυρία καμαέβερτ για τα 6 ή 10 εκατομμύρια. Θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε αυτό, να αποφασίσουμε τι είναι καλύτερο. Όχι όμως σε επίπεδο περιεχομένου δεν θέλουμε αυτόν τον προπολογισμό. Και αυτό ισχύει και για τι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Να αναφέρω ένα από τα πολιτικά προγράμματα των Πρασίνων. Η ιδέα ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ έρευνα και έρευνα για το πώς μπορούμε να ε, προωθήσουμε την επικοινομορφία σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Έχουμε διάφορες δυνατότητες από την κοινότητα του διαδικτύου και θεωρώ ότι θα πρέπει πραγματικά να επενδύσουμε σε πιο πολύ έρευνα στον κλάδο αυτό για να υπάρξουν πιο πολλά μοντέλα χρηματοδότησης ε, πολιτισμικής ποικιλομορφία στην ψηφιακή εποχή. Ελπίζω να υπάρξει υποστήριξη για την στρατηγική τώρα, για την επικοινωνία που ανέφερε ο Μόρτεν. Είμαι έξαλλη τον ακούω αυτά που μας είπε για παράδειγμα η κυρία Ρέντινγκ την τελευταία φορά που της μιλήσαμε απέριψε την όλη ιδέα των ε, τηλεοπτικών δικτύων. Το να περάσουμε τώρα στο, στα φυλάδια σε μια εποχή όπως η σημερινή είναι κάτι το οποίο δεν πείθει καθόλου. Και αυτό που πρέπει να αναπτύξουμε τα αρδιοφωνικά και τα λεοπτικά δίκτυα θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη επιρροή. Ιδιαίτερα για τη Γερμανία, τις σκανδιναβικές ε, και τις βόρειες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή γιατί υπάρχει καλή κάλυψη. Η Επιτροπή Πολιτισμού δεν μπορεί να δεχτεί αυτά που κάνει. Δεν μπορεί να δεχτεί το ότι δεν ακολουθεί τις απαιτήσει που έχουμε θέσει. Και προφανώς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να είμαστε ξεκάθαροι για τα συμφέροντά μας και να δείξουμε στην Επιτροπή Ρέντινγκ ότι δεν θα μπορέσουμε να αποδεχτούμε άλλο αυτά που κάνει ή μάλλον αυτά που δεν κάνει. Κύριε Χόνιμπολ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι για την ε, διαβίου μάθηση και γενικά για τις εταιρικέ σχέσεις ε, για την γνώση. Πολύ καλή ιδέα τώρα για τον αθλητισμό. Αν μπορούσαμε να ζητήσουμε πραγματικά αυτά τα οποία θέλουμε να ζητήσουμε, περιμένοντας να λάβουμε ένα λογικό ποσό, αξίζει να το δοκιμάσουμε. Το σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε. Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική για την επικοινωνία. Δεν ξέρω αν θα το συζητήσουμε αυτό και στη συνάντηση των συντονιστών. Πάντως, γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι ε, ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή απλώς δεν λειτουργεί. Και από τη σκοπιά της Βρετανίας θεωρώ ότι είναι ο χειρότερος δυνατός τρόπος για να διεξάγει κανείς μια πολιτική επικοινωνία. Αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να ενημερώνουμε τελικά τον Ευρωπαίο πολίτη για το τι γίνεται εδώ, και αν θέλουμε πραγματικά να προσελκύσουμε και να αφυπνίσουμε τους πολίτες, προφανώς δεν το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Δεν το έχουμε πετύχει αυτό και τα πράγματα επιδεινώνται τελικά, να βελτιώνονται. Συνεπώς, νομίζω ότι απαιτείται μία κάποια στρατηγική τουλάχιστον, μία στρατηγική όμως αποτελεσματική, μία στρατηγική που να ενημερώνει πραγματικά τους πολίτες για το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πολιτική που θα βοηθά τους πολίτες να καταλάβουν ότι κάνουμε μια καλή δουλειά, ότι έχουμε μια δημιουργική στάση, ότι εξ ονόματό του ουσιαστικά και για αυτού εργαζόμαστε εδώ πέρα. Και θεωρώ ότι ακόμα και αυτό το βασικό μήνυμα δεν έχει περάσει. Λοιπόν, πρέπει να μα απασχολήσει σοβαρά η πολιτική αυτή. Χρειαζόμαστε βέβαια τον απαραίτητο χρόνο για να την καταρτήσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριο Λόκεγκάρτ έθεσε το ζήτημα αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να λάβουμε αυτή τη στιγμή μια τελική απόφαση. Οι επιμέρου πολιτικέ ομάδε χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα περισσότερο. Ευχαριστώ. Ε, ναι, αλλά σας είπα και ποιες είναι οι προθεσμίες, εντάξει. Ας το έχετε αυτό κατά νου. Η κυρία Σάκε, σας ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τις αρχικές σας σκέψεις για τον προπολογισμό. Πρόκειται για περίπλοκο ζήτημα και ως Ολλανδέζα γνωρίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να κάνουμε πιο πολλά με πιο λίγα χρήματα. θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, ιδιαίτερα δεδομένων των ε, δυνατοτήτων που μας δίνουν ε, τα νέα μέσα για την ε, επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς απαραίτητα μετακίνηση, το οποίο κοστίζει. Θα ήθελα επίσης να μοιραστώ μαζί σας μία ιδέα ενός πληροτικού προγράμματος εξ ονόματος της ομάδας. Έγινε πρόσφατα ακρόαση που εξέτασε θέματα ευκαιριών και εκπαίδευσης για τους νέους και η Χιλέν Δερβέν, η οποία είναι ιδρύτρια των ε, σχολείων Κυριακού, που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε παιδιά από περιβάλλοντα χωρίς πολλές ευκαιρίες προκειμένου να ε, μπορούν τα Σαββατοκύριακα να εκπαιδεύονται σε τομείς όπως ε, πυροσβέστες, ε, γιατροί και το καθεξής. Αυτό το πληθυντικό πρόγραμμα προτείνει να χορηγηθούν χρήματα για project όπως ευρωπαϊκά ευρωπαϊκές κατασκηνώσεις, θερινές κατασκηνώσεις, με το ίδιο σχέδιο για να αυξηθούν οι διεθνείς ικανότητες, να αυξηθεί η κινητικότητα. Αν θέλετε άλλες πληροφορίες, ευχαρίστω να σας τις δώσω. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι η γραμμή αυτή του προϋπολογισμού που είναι τόσο σημαντική θα λάβει την υποστήριξή μας. Κυρία Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον εισηγητή. Τρία πράγματα θα θέλω να πω. Πρώτον, σωστό τα όσα προτείνει για τον ε, προϋπολογισμό, για τις ε, προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να τεθούν και για τις αυξήσεις που θα πρέπει να έχουμε στις συγκεκριμένες προτεραιότητες καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι ο πολιτισμό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα είναι όμω ότι ο προπολογισμό από ό,τι φαίνεται παραμένει στάσιμο και τίποτα δεν αλλάζει. Όταν περνάμε μάλιστα στα πολιετή προγράμματα, εκεί πέρα βλέπουμε ότι το 2012 θα αποτελέσει έτος ενδεικτικό για τα μελλοντικά έτη. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να πετύχουμε περισσότερο το 2012 γιατί αυτό θα σημάνει και τη γενικότερη τάση που θα επικρατήσει στο μέλλον. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μειωθούν τα κονδύλια για τον πολιτισμό. Είναι πολύ κρίσιμα αυτά λοιπόν τα οποία πρέπει να αποφασιστούν. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, έχω την εντύπωση Ίσως ο συνάδελφος να μπορέσει να με διαφωτίσει. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε μία μεσογειακή πολιτική, πολύ σημαντική για τη συνεργασία ανάμεσα στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όχι μόνο μεταξύ μόνα αλλά και τρίτων χωρών. Μα ακόμα και σε αυτά τα προγράμματα βλέπω τελικά ότι υπάρχει μια σημαντική περικοπή του προπολογισμού. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια για να αυξηθεί και αυτή η συνεργασία και να αυξηθεί και η κινητικότητα των νέων. Ξέρετε ότι αναφερόμαστε όλο και περισσότερο στη διαβίου μάθηση και πώς αυτή συνδέεται με την κινητικότητα, μα νομίζω ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι θα υπάρχει τροποποίηση όσον αφορά τα προγράμματα κινητικότητα στο μέλλον και όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται τα προγράμματα αυτά να ενισχυθούν αν δεν αυξηθούν και τα κονδύλια. Και αύξηση τα κονδύλια εγώ δεν βλέπω. Ξέρετε επίση ότι ε, η στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάπω περίεργη όσον αφορά το θέμα τη επικοινωνία. Στο παρελθόν, από θεωρητική πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρούσε σε παρουσίες επικοινωνικών προγραμμάτων, η οποία ήταν καταπληκτική. Στη συνέχεια όμω βλέπουμε ότι μειώνεται χρηματοδότηση. Δεν νομίζετε εδώ πέρα ότι υπάρχει πραγματικά μία αντίφαση. Προσπαθούμε απλώς να δώσουμε εξωτερικά μία θετική, ε, ωρεοποιημένη εικόνα των πραγμάτων. Το ζήτημα αυτό το είχα θέσει και σε παλαιότερη ακρόση που είχαμε με τον Επίτροπο και νομίζω ότι θα πρέπει να τεθεί εκ νέου. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφερόμενη σε επικοινωνία, να θέλει απλώ να κάνει μια κάποια πολιτική δήλωση και να μην έχει τελικά μια έμπρακτη πρόθεση να προχωρήσει σε κάτι πιο απτό. Ας ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την ουσία των θεσμικών οργάνων και όχι τόσο πολύ με τον τρόπο που αυτά ε, παρουσιάζονται προς τα έξω. Βλέπουμε επίσης ε, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για το 2013 και για την συνέχεια. Θεωρώ εδώ πέρα πάλι ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση όσον αφορά τόσο τις πληρωμές και την άλλη υποχρεώσεων. Πώ κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία επιπλέον παρατηρήση επιτρέψτε μου. Η στρατηγική για την επικοινωνία. Θα με ενδιαφέρει να ξέρω αν ε, μπορεί να ε, εκτιμηθεί η αποδοτικότητα, γιατί στην παρούσα φάση διακυβεύεται έντονα η ευρωπαϊκή ιδέα και κάθε ε, ραδιοφωνική ώρα, κάθε εκπομπή για την Ελλάδα καταστρέφει πάρα πολλά αυτά που, που αναπτύξαμε επί τόπου. Και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, το θέτω ως θέμα, ίσως για την Επιτροπή, για την εργασία μας, να, δώσουμε, να αναθέσουμε την εξαγωγή μιας μελέτης για την ε, αποτελεσματικότητα της στρατηγικής επικοινωνίας. Μιλάμε για την αποδοτικότητα της επικοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό θα μας ωφελούσε. Ποιος μικροφώνου, η Πρόεδρος. Ο κ. Λόκιγκαρτ έχει το λόγο και μετά μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συγχωρείτε. Πολύ σύντομα. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είμαστε σαφώς υπέρ της πρόθεσής σας αυτής να υπάρχουν πιο συγκεκριμένε προτεραιότητες και χαιρόμαστε πάρα πολύ με την έμφαση που δίδεται στην διαβίου μάθηση και στον αθλητισμό. Ως προς τον αθλητισμό να πω κάτι ακόμα για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει νέα κονδύλια για το 2012. Αυτό μας ρωτήσατε. Κοιτάξτε, να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Το 2011 είναι το τελευταίο έτος της προπαρασκευαστικής δράσης. Σύμφωνα λοιπόν με τον χρηματοπιστωτικό κανονισμό, είτε πρέπει να προτείνει ένα νέο πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νομική βάση για περαιτέρω χρηματοδότηση και κάτι τέτοιο ξέρετε ότι εμείς το κάνουμε για την περίοδο μετά το 2013 Σαφώς βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί ακόμα να προτείνει ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα για τον αθλητισμό. Και όπως σας είπα, είμαστε σαφώς υπέρ του να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό ανάμεσα στο 2011 και το 2014. Ετέθηκε ένα ερώτημα για τον προπολογισμό όσον αφορά τους νέους. Για ποιο λόγο δεν αυξάνεται περισσότερο, μας ρωτήσατε. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η βάση της εργασίας μας είναι το ο πολιετής προγραμματισμός για τα προγράμματά μας. Και όπως και στα παρελθόντα έτη, ο προπολογισμό για τους νέους είχε λάβει περισσότερα χρήματα χάρη στις δικές σας προσπάθειες. Διακινδυνεύσαμε ακόμα και με μείωση του προπολογισμού για το 2012 για την νεολαία. Αν είχαμε ακολουθήσει απλώς τον πολιετή προγραμματισμό, θα είχαμε δει τότε σαφώ μία μείωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταυτού πρόσθεσε νέα κονδύλια στην εν λόγω γραμμή προπολογισμού ώστε να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει αύξηση του προπολογισμού για τα προγράμματα νεολαίας για το 2012. Προβλέπεται λοιπόν από το 2011 προς το 2012 μία αύξηση, μολονότι δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο στον πολιετή προγραμματισμό. Εν κατακλείδη λοιπόν είμαστε υπέρ της δικής σας ε, εστίασης σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Θα εξετάσουμε και άλλες ενδεχόμενες προτάσεις και τροπολογίες που θα έρθουν από εσά και θα κάνουμε βέβαια και εμείς κάποιες ε, παρατηρήσεις τεχνικής φύσεως στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Είναι κανείς από την Διεύθυνση Επικοινωνίας ε, της Επιτροπής. Α, κρυβόσαστε. Α, μάλιστα, βεβαίως, βεβαίως. Σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ συνάντηση με τον ε, κύριο Λόκουγκάρτ και παρουσιάσαμε την άποψή μας για διάφορα από τα θέματα που παρουσίασε ο κύριος Λόκεγκάρτ. Νομίζω ότι το ερώτημα για την ε, περίοδο αυτή τα συζητήσαμε και πέρσι αυτά. Παρουσιάσαμε τη σχετική τη σχετική παρουσίαση, τη σχετική έκθεση και υπήρξε η ιδέα ότι αυτά ήταν εικονοποιητικά για την Επιτροπή σας σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μας για την ε, επικοινωνία. Η κυρία Ρέντινγκ ήρθε στην Επιτροπή και μας ε, παρουσίασε την προσέγγιση αυτή στην επικοινωνία. Λάβαμε λοιπόν τα σχόλια αυτά και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, κύριε Λόκεγκάρτ. Ευχαριστώ. Ακούστε. Λίγε παρατηρήσει έχω να κάνω σε σχέση με αυτό που υπόθηκαν για τον αθλητισμό. Συμφωνώ πλήρω ότι ίσω τα 6 εκατομμύρια να μην είναι το σωστό ποσό. Μπορούμε να το συζητήσουμε, σα το είπα και πριν. Αλλά θα πρέπει να μα εξηγήσει και η Κομισιόν. Νομίζω ότι τα 3 εκατομμύρια που έχουμε με τα 6 εκατομμύρια ή τα 5 εκατομμύρια δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Μιλάμε για δύο χρόνια, για τρία χρόνια. Δεν ήταν σωστή η διαίρεση που κάνατε, αλλά τέλος πάντων. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ίσως αυτό το νούμερο δεν είναι αρκετά υψηλό. Και θα πρέπει ίσως αυτό να το ξεκαθαρίσουμε στις διαπραγματεύσεις. Αλλά μην διστάσετε, πείτε 10, 20, 30, κανένα πρόβλημα από δική μου πλευράς. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τα σχόλια για τις πολιτικές επικοινωνίας. Εγώ είχα διαφορετική άποψη, δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, αλλά συμφωνώ ότι θα πρέπει να το συστήσουν και ομάδες. Καλό θα ήταν πάντως, το συντομότερο δυνατό, οι συντονιστές των επιτροπών ε, να τα συζητήσουν σε μια συνεδρίαση και μετά να κάνω και εγώ τις προτάσεις μου. Επίσης μίλησαμε για το χρόνο. Εδώ και 1,5 χρόνο επεξεργαζόμαστε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι όλοι, τουλάχιστον έτσι νομίζω, ψηφίσατε υπέρ της έκθεσής μου, όπου περιλάμβανε 50 διαφορετικές ε, υποδείξεις και προτάσεις. Καμία όμως δεν εισακούστηκε, τις ψηφίσαμε όμως. Τελικά θέλουμε απλά να συζητάμε την επικοινωνία και την πολιτική αυτή. Φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να είμαστε βέβαια λογικοί, αλλά να δούμε και κάποια πράγματα, κάποια πράξεις, όχι μόνο λόγια. Ψηφίσαμε αυτή την έκθεση και αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαφετηρίας. πάντως από ό,τι θυμάμαι για αρκετούς μήνες διαπραγματευόμαστε την έκθεσή μου. Άρα νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το χρόνο πλέον φτάνουμε ε, στο τέλος της διορίας. Γι' αυτό είπα αυτά που είπα. Πάντω θέλω να σα ευχαριστήσω για τα σχόλια και για την υποστήριξή σα ό,τι αφορά τα διάφορα κονδύλια του προπολογισμού. Να σας πω ενημερωτικά ότι η κατάθεση των τροπολογιών ε, μπορεί να γίνει μέχρι τις 27 Ιουνίου. 27 Ιουνίου η λίγη προθεσμία λοιπόν κατάθεση τροπολογιών όπως είπε και η Πρόεδρος και στις 14 Ιουλίου έχουμε μια άλλη προθεσμία. Προσβλέπω πάντως, ε, αναμένω τέλος πάντων με της της διαπραγματεύσεις. You all for being here. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είσαστε εδώ πέρα και έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ. Ω, Χριστέ μου. It was my wishing. Ναι, ήταν ευσεβής πόθος ίσως. Ζητώ συγγνώμη από το Σαντιάγκο. Το θέμα είναι τόσο σημαντικό. Ο αθλητισμός είναι τόσο σημαντικός. Σου δίνει το λόγο. Ευχαριστώ, Δόρη. Σε συγχωρώ. Δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα. Ήδη πάντως είχαμε κάνει μια πρώτη ανταλλαγή εντυπώσεων, ιδιαίτερα ευρεία. Και πολύ ενδιαφέρουσα ήταν επίσης η συζήτηση που είχαμε, αλλά και οι ερωτήσεις ε, και οι παρεμβάσεις των συναδέλφων. Ουσιαστικά έχω ολοκληρώσει την τελική έκθεση. Το μόνο που λείπει είναι να ολοκληρώσω τις προσαρμογές ε, στο περιορισμένο χώρο που έχω στη διάθεσή μου. Δεν μπορεί να υπερβαίνει δηλαδή μια συγκεκριμένη έκταση αυτή η έκθεση, άρα πρέπει να την ψαλιδίσω λίγο. Νομίζω θα τη συζητήσουμε στη συνεδρίασή μας τον Ιούλιο, οπότε αυτό που μπορώ τώρα να κάνω είναι να σας εξηγήσω λίγο τις αντρές γραμμές. Όταν όμως συζητήσουμε την έκθεση ε, τον Ιούνιο. Δηλαδή, όταν αποφασιστεί η συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε θα τα πούμε επί της ουσίας. Δύο είναι τα βασικά σύνορα. Το πρώτο είναι η αρχή της επικουρικότητας ε, των κρατών μελών που πρέπει να την εφαρμόζουμε, να την τηρούμε και το δεύτερο είναι η ιδιαιτερότητα του αθλητισμού. Δηλαδή η δύναμη που έχουν οι διάφορες ομοσπονδίες για παράδειγμα. Η ιδιαιτερότητα αυτή όμως δεν θα πρέπει να αποτελέσει γενικό κανόνα. Είναι κάτι που πρέπει να μελετάτε κατά περίπτωση. Επαναλαμβάνω, θα συνοψίσω κάποιες βασικές ιδέες και εν συνεχεία ίσως καλό θα ήταν οι συνάδελφοι να μου θέσουν τα ερωτήματά τους και θα προσπαθήσω να απαντήσω στο σύνολο. Και στην έκθεση βέβαια θα περιορίσω σίγουρα το κείμενο και θα προσπαθήσω να είμαστε δυνατόν πιο πλήρη. Ποιο είναι το βασικό λειτουργήμα του αθλητισμού. Είναι η ενίσχυση τη άσκηση τη άθληση στα σχολεία, στα διάφορα ε, ιδρύματα και βέβαια ε, την ε, ένταξη. Φυσικά τα άτομα με αναπηρία πώς θα έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό. Έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες και ιδέες για αυτό το θέμα. Ανάπτυξη επίσης του γυναικείου αθλητισμού ιδίως ό,τι αφορά την υποεκπροσώπηση των γυναικών ε, σε υψηλά αξιώματα, καταπολέμηση επίσης της φαρμακοδιέγερσης. Υπάρχει μια πρόταση που ίσως είναι λίγο παρακινδυνευμένη, δηλαδή η δημιουργία μιας ε, αντιπροσωπείας ε, του ΚΑΣ, του Αθλητικού Δικαστήριου, του στο Λουξεμβούργο της Βρυξέλλες. Καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα ε, είναι επίσης μια πρόταση, καθώς επίσης και ε, η δημιουργία ενός καταλόγου με hooligans που θα τους απαγορεύεται είσοδος σε αγωνιστικούς χώρους, σε αθλητικές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις και βέβαια στήριξη της εκπαίδευσης ε, των αθλητών, διπλή σταδιοδρομή, είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με συγκεκριμένες προτάσεις κάποια ε, συνοδευτικά προγράμματα, διευκολύνσεις ε, για την επαγγελματική του ε, σταδιοδρομία, για τις πανεπιστημιακές σπουδές και ούτω καθεξής. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά και συγκεκριμένα ότι πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αθλητισμού και περιβάλλοντος. Σκι, γκολφ. Πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία. Σε ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση, πρέπει να τονίσουμε τον εθελοντισμό και τη σημασία ότι υπάρχουν 35 εκατομμύρια Ευρωπαίων εθελοντών και χωρίς αυτούς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθεί το αθλητικό μας σύστημα και ιδίως ε, ό,τι αφορά ε, τον αθλητισμό για όλους, τον μη επαγγελματικό αθλητισμό και επίσης θα πρέπει να δούμε για τα σωματεία και τις ενώσεις ε, τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Βέβαια, εναπόκειται στα κράτη-μέλη αυτό, αλλά ουσιαστικά απευθύνουμε άγκληση στα κράτη-μέλη να στηρίξουν με ειδική φορολογία τις διάφορες ενώσεις ε, και σωματεία. Δεν μιλάω για τα επαγγελματικά σωματεία, μιλάω για τους ε, ερασιτεχνικούς συλλόγους, τα ερασιτεχνικά σώματα και συνεργασία με την WADA, τον Οργανισμό για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ. Επίσης έγινε λόγος ε, για την ρύθμιση των, των στοιχημάτων. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι μια βασική αρχή θα ήταν να αναγνωρίσουμε την πνευματική ιδιοκτησία, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των οργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να αποφύγουμε τα πρακτορία στοιχημάτων να μπορούν να στοιχηματίζουν επί παντός επιστήτου. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια ρύθμιση του στοιχηματισμού. Επίσης, ό,τι αφορά την πώληση των κεντρικών τηλεοπτικών ε, δικαιωμάτων, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και βέβαια και στη χώρα μου είναι ένα ζήτημα πολύ ε, σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τώρα την οργάνωση του αθλητισμού, θα πρέπει να στηρίξουμε σαφώ το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στι ομοσπονδίε, ε, στα σωματεία και στου εθελοντέ. Το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο δεν έχει καμία σχέση με το αμερικανικό. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα. Πρέπει νομίζω να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο. Επίση, ανάγκη καλή διακυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς σεβόμαστε με την αυτονομία των ομοσπονδιών, αλλά θα πρέπει ω αντάλλαγμα να ζητήσουμε από αυτέ πραγματική δημοκρατία όλοι οι stakeholders για να το πω στα αγγλικά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οι εμπλεκόμενοι όσοι έχουν λόγο θα πρέπει να εκπροσωπούνται στις αθλητικές διοργανώσεις και φορείς να υπάρχει πραγματική δημοκρατία πραγματική διαφάνεια. Επίση, Επίσης η ακαιρεότητα των αθλητικών διοργανώσεων. Θα πρότεινα τα κράτη να ανακηρύξουν ως αξιόπινη, ποινικά αξιόπινη πράξη ε, οποιαδήποτε ε, παρέμβαση στις διοργανώσεις θα πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα, να, οριστεί ένα ποινικό αδίκημα. Ρύθμιση επίσης ε, των δραστηριοτήτων των μάνατζερ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει και με τις ε, μετεγγραφές ε, των παικτών. Η ΦΥΒΑ ζητά απορρίθμιση, εγώ ζητώ το αντίθετο πρέπει να γίνουν ίσως κάποιες ε, ε, τροποποίησεις, πρέπει να έχουν κάνει πανεπιστημιακές σπουδές αυτοί οι μάνατζερ και να έχουν ε, την έδρα τους σε μια χώρα της Ένωσης και όχι σε ένα φορολογικό παράδεισο. Και επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί μια λίστα, ένας κατάλογος των παικτών που εκπροσωπούν αυτοί οι μάνατζερ και τι σχέσεις έχουν με αυτούς. Και κυρίως θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Υπάρχει ένα νέο κεφάλαιο που νομίζω ότι είναι σημαντικό και συγκεκριμένα συνεργασία με τρίτες χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε σε όλες τις συμφωνίες συνεργασίας να συζητούν διάφορα προβλήματα όπως είναι η πειρατεία, η εκμετάλλευση ανήλικων αθλητών, παράνομος στοιχηματισμός, γιατί πολλά πρακτορία στοιχημάτων έχουν την έδρα τους σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα ήταν δυνατό ενδεχομένως να στηριχθούν κάποιες πολιτικές ανάπτυξης μέσω του αθλητισμού, βελτίωση της υγείας, ένταξη κοινωνική ένταξη, ένταξη της ε, γυναίκας, ε, μιλάμε για χώρες του κόσμου και ούτω καθεξής. Τέλος, κάτι που έχω ξαναπεί, ευρωπαϊκή ταυτότητα του αθλητισμού. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το άρθρο 165 Τη συνθήκη της Λισαβόνας κάνει λόγο για την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Δεν είναι δηλαδή δική μου εφεύρεση. Εγώ προτείνω τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής ημέρας αθλητισμού να στηρίξουμε τον αθλητισμό να έχουμε ένα χάρτη των παραδοσιακών αθλημάτων και θα μπορούσαμε ίσως να δημιουργήσουμε και ένα φεστιβάλ παραδοσιακών αθλημάτων στα μεγάλα αθλητικά ε, γεγονότα να κυματίζει η ευρωπαϊκή σημαία επίσης, όχι μόνο η χώρα ε, της χώρας της διοργανώτριας και ένα ε, πρόγραμμα κινητικότητα σε ένα είδους ε, Προγράμματο Εράσμου, πιλωτικό πρόγραμμα, το είπα και πριν όταν μιλήσαμε για τον προπολογισμό, που νομίζω ότι θα μπορούσε να το στηρίξει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων της Επιτροπής μας. Βέβαια θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους, να ζητήσω και να προσφέρω τη συνεργασία μου προς όλους τους κοιόδες εισηγητές των διαφορετικών πολιτικών ομάδων αλλά και των διαφορετικών επιτροπών που θα γνωμοδοτήσουν και φυσικά είμαι ανοιχτός και στη συνεργασία αυτή και σε οποιαδήποτε ερώτηση. Θα μπορούσα να ε, μακρηγορήσω, να επεκταθώ ακόμη περισσότερο, αλλά ήθελα να σας διαγραφήσω τις βασικές γραμμές της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Σαντιάκο. Και τώρα ζητούν πέντε συνάδελφοι τον λόγο. Δεν θα ολοκληρώσουμε γρήγορα τελικά σήμερα. Ο κύριος Μπελέτα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ συνοπτικός και ακριβής τρία σύντομα στοιχεία, πολύ συγκεκριμένα. Καταρχάς για την ε, την και τους ε, μάνατζερ των ε, παίκτων. Όχι προς αντιγραφή της πρότασης της FIFA και για να παρουσιάσουμε ένα εναλλακτικό μοντέλο. και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να το σχολιάσει αυτό γιατί σήμερα αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες ε, υπάρχει διάλογος μεταξύ της Κομισιόν και των παικτών και των διαφόρων ομοσπονδιών. Είναι σημαντικό λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη ε, τις προτάσεις που τίθενται και σε αυτό το πλαίσιο προκειμένου να προσπαθήσουμε να, την, ε, να τις συμπεριλάβουμε και αυτές. Κατά δεύτερον, Αναφέρατε, Πρόεδρε, το ιδιαίτερο καθεστώς των ε, λεσκών αθλητισμού. Το συζητήσαμε και πριν από κάποια χρόνια το θέμα αυτό. Μιλήσαμε για τα δικαιώματα τέτοια ε, λέσχης για να, έχουν, ε, να έχει ιδιαίτερο καθεστώς κοινωνική ασφάλεια κτλ. Αλλά μιλήσαμε και για το θέμα των υποχρεώσεων, των κοινωνικών υποχρεώσεων καλή ιδέα θα ήταν ίσως να προσπαθήσουμε όχι να εναρμονίσουμε, αλλά να καταλήξουμε σε κάποιες ε, καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά τις αθλητικές λέσχες. Τελευταίο στοιχείο, Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σημαντικό, αφορά και πάλι τα θέματα ακεραιότητας και συγκεκριμένου χαρακτήρα, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό στην έκθεση για την καλή διαχείριση κάποιων τέτοιων ε, ενώσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την FIFA, γιατί πολλά συμβαίνουν στο πλαίσιο της FIFA τις τελευταίες εβδομάδες και θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής απάντηση. Και ο καλύτερος τρόπος είναι η έκθεση αυτή. Νομίζω ότι η εκλογή του νέου Προέδρου καλό θα ήταν να μην έχει γίνει. Και τώρα η FIFA έχει συστήσει ένα συμβούλιο σοφών, όπως το ονομάζει, για να ξεκινήσει μία ανεξάρτητη έρευνα. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όταν μιλάμε για το δικαίωμα τέτοιων ενώσεων να έχουν ξεχωριστή μεταχείριση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά που προτείνει η FIFA και νομίζω ότι είναι σαφής η αντίδραση της Επιτροπής. Συμφωνούμε με την ειδική μεταχείριση των ε, διοικητικών όργανων αρκεί να υπάρχει σεβασμό στην ακαιρεότητα και να υπάρχει συγκεκριμένη διαφάνεια. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό στη FIFA και ίσως θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά ανεξάρτητη έρευνα γιατί όλοι οι φίλαθλοι έχουν δικαίωμα σε μια ανεξάρτητη τέτοια μελέτη. Κυρία Χάνιμπαρ. Σας ευχαριστώ. Μία δήλωση θα ήθελα να σας διαβάσω από τον κύριο Ιβάν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι εδώ πέρα σήμερα, λυπάται που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, μου ζήτησε όμως να στη διαβάσω και θα ήθελα να κάνω πρώτα κάποιες παρατηρήσεις. Συμφωνώ μετά τα όσα είπε ο κύριος Μπέλετ για, τη FIFA. Θα είναι πολύ καλό αυτό και να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Θα ήθελα να συμφωνήσω και με τον εισηγητή στα όσα είπε για τις γυναίκες. Όντως υποεκπροσωπούνται και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λέμε στην έκθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την αναφορά και να σας διαβάσω και τη δήλωση. Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοιε αναγνώσει εδώ πέρα. Δώστε τη δήλωση στον κύριο Φίσα για να τη λάβει υπόψη του. Δεν νομίζω ότι μπορείτε αυτή τη στιγμή να παίρνετε το λόγο και να διαβάζετε δηλώσει. Α ήταν εδώ πέρα για να τη διαβάσει. Είστε πολύ καλοί μαζί του, αλλά δώστε το. Δώστε τη δήλωση αυτή στον κύριο Φίσα και θα τη λάβει υπόψη του. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Τέρο, κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα ως ε, αθλητής που αναφερόμαστε σε, ε, σε τέτοια παραπτώματα σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Η καταπολέμηση του ντόπινγκ είναι πολύ σημαντική. Και στη Φιλανδία επίσης υπάρχουν τέτοιοι εγκληματίες οι οποίοι έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τον αθλητισμό προσδίδοντας κακή φήμη και αυτό παρατηρήθηκε και πριν από κάποια χρόνια στο φιλανδικό baseball. Είναι πολύ σημαντικό να απαλληφθεί η διαφθορά στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός ε, περιλαμβάνει μεγάλο, μεγάλα χρηματικά ποσά, 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ διαβάζουμε στην έκθεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ως οικονομικό μέγεθος, αλλά και ως συμβολικό ποσό, γιατί οι νέοι σέβονται τους αθλητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αποστέλλεται τέτοια μηνύματα από τον κόσμο του αθλητισμού, γιατί οι άνθρωποι, αυτά, οι άνθρωποι αυτοί είναι συχνά τα είδωλα των νέων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή. Ευχαριστώ, κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Βασικά ρωτήσεις να κάνω προς τον εισηγητή σας. Ευχαριστούμε για την εισαγωγή. Μιλήσατε για το δικαστήριο για το ντόπινγκ. Τι εννοείται. Ότι η αρμοδιότητα για τον ντόπινγκ θα φύγει, θα μεταφερθεί αλλού. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τους χούλιγκαν, θα ήθελα να μου δώσετε πιο πολλές πληροφορίες, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το σημείο αυτό. Και τελευταία ερώτηση. Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται καταπηγόντως μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη διαχείριση της FIFA, γιατί έτσι επηρεάζεται η φήμη όλου του αθλητισμού. Θα πρέπει φυσικά να υπάρξει ανεξάρτητη έρευνα και θα πρέπει να διασφαλίσουμε κάτι να γίνει με το έργο αυτό, με το αποτέλεσμα της ανεξάρτητης έρευνας, να μην χαθεί σε κάποιο σιρτάρι. Ευχαριστώ κύριε Μπόρις Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο. Ουσιαστικά τα ανέφερε όλα. κατάφερε να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία μιας πολύ σύνθετης κατάστασης. Η πολιτική θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Ταμείο, από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, να υπάρξει ένα μέσο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ένα τμήμα των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν θα πανάτε μόνο για δρόμους, αλλά και για αθλητικές εγκαταστάσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην παρούσα φάση. Και κάτι άλλο, φυσικά είναι πολύ εκτενής η έκθεση. Θα ήθελα όμως να προσθέσουμε άλλο ένα στοιχείο, ότι ο αθλητισμός και ότι οι βασικέ δεξιότητε στον τομέα του αθλητισμού θα πρέπει να λεφτούν υπόψη. Μιλήσαμε για τι βασικέ δεξιότητε και νομίζω ότι ο τομέας αυτός θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Γιατί αποτελεί ένα πόρο εν δυνάμει. Θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν και οι εθνικές αρχές σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της καινοτομία και των ε, μέσων προκειμένου να έχουν πιο, πολύ, πιο πολλές καλές συνθήκες οι νέοι στην εθνική πραγματικότητα, η αίμα. Σας ευχαριστούμε, Σαντιάγκο, για τη δουλειά σας και για την, ε, το ακούραστο έργο σας. Θα ήθελα κάτι να σχολιάσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εργάζεται εκεί που έχει προσθεθέμενη αξία. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να ε, ενισχύσουμε τον αθλητισμό. Συζητάμε για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Πώς μπορούμε να κοιτάξουμε το θέμα της χρηματοδότησης του αθλητισμού. Και είναι σαφές ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, τη χρηματοδότηση που υπάρχει και τα μοντέλα που υφίστανται. Θα πρέπει να προσέξουμε γιατί οι ροές που υπάρχουν θα πρέπει να τις προστατεύσουμε. Μπορεί να μην χρειαζόμαστε νέα μοντέλα, αλλά χρειάζεται σύμβορα ε, διαφάνεια και θα πρέπει να προωθηθεί. Επίσης μιλήσατε και για την αυτονομία των οργανώσεων αυτών, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να εκπροσωπούνται στις συναντήσει αυτές. Αυτό είναι πασιφανές, θεωρώ υποστηρίζω την ιδέα του αθλητισμού, του εράσμους αθλητισμού. Δεν είμαι τόσο υπέρ μιας ευρωπαϊκής σημαία σε όλες τις εκδηλώσεις. Αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να επιβληθεί. Μπορεί να το θέλει, μπορεί να περάσει τελικά αυθόρμητα. Και επίσης δεν μπορούμε να επιβάλλουμε επιπλέον γραφειοκρατία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ανάπτυξη του αθλητισμού και αυτό θα γίνει από κάτω προς τα πάνω. Ο Μάρκος Κουρία. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ε, έκθεση του Σαντιάγκο είναι πολύ καλή, πολύ πλήρης, περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάποια επιμέρους σημεία. Θυμάμαι ότι τα είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Το να δημιουργήσουμε το θεσμό της Ευρωπαϊκής πρωτεύουσα Αθλητισμού. Ενδεχομένω αυτό να αποτελέσει μια κάποια θεσμική καινοτομία την οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και να αναφέρουμε σε αυτή την έκθεση. Δεύτερον, ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Σαντιάγκο ήδη και το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο συγκεκριμένα να ασχοληθούμε περισσότερο με τη θέση των γυναικών στον αθλητισμό. Κάθε φορά που μιλάμε για συνεργασία με τρίτες χώρες, θα μπορούσαμε μέσω του αθλητισμού να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών σε χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά οι οποίες έχουν μια κάποια αθλητική παράδοση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές στην έκθεση και θα πρέπει να σε απασχολήσει ιδίως από τα προγράμματα που θα έχουμε, στα προγράμματα που θα έχουμε από το 2012 και μετά. Επίσης, πολύ συχνά οι πολίτες δεν μπορούν να ασχοληθούν με αθλήματα γιατί λείπει η βασική υποδομή. Ίσως λοιπόν να μπορούσαμε να αναφερθούμε σε κάποια προγράμματα εξοπλισμού κάποιων αθλητικών κέντρων, μια κάποια ενίσχυση που θα μπορούσε να δοθεί σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να υπάρχει αυτή η υποδομή. Δεν αναφέρομαι σε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις προφανώς. Ίσως θα μπορούσαμε όμως μέσω μιας κάποιας χρηματοδότησης να βοηθήσουμε πολλούς νέους ή και μη νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό περισσότερο. Η έκθεση λοιπόν του Σαντιάκο Φίσας θα πρέπει να αναφερθεί και σε αυτό. Δηλαδή να πούμε ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να είναι διάχυτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσβάσιμο σε όλους. Η κυρία Κώστα, πολύ σύντομα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή μας, τον Σαντιάγκο Φίσας. Τρεις παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Πρώτον, χαίρομαι πολύ που είχε ασχοληθεί πάρα πολύ σε μια σύντομη ουσιαστικά έκθεση, προσπαθώντας να καλύψει πολλές διαφορετικές πτυχές του ζητήματος. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση για τον αθλητισμό. Ενδεχομένω να πρέπει να καταφύγουμε και σε κάποιε συνέργειε προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε την ευκταία αυτή χρηματοδότηση. Να ασχοληθούμε περισσότερο και με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών μέσω του αθλητισμού. Ξέρετε ότι ο αθλητισμό δεν χρηματοδοτείται επαρκώ και ακόμα λιγότερο βέβαια ο αθλητισμό για τι γυναίκε. Επομένω κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Μία από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι η διάχυση του αθλητισμού, η διάδοση του αθλητισμού, η δημιουργία καλύτερων υποδομών προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Για να τα πετύχουμε λοιπόν αυτά, ίσως θα πρέπει να επινοήσουμε και κάποιες προδιαγραφές για τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές, προκειμένου να γνωρίζουν τι επενδύσεις θα πρέπει να κάνουν στο τομέα του αθλητισμού. Κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνει ο αθλητισμός πολύ πιο προσβάσιμος στις τοπικές κοινωνίες, στα πανεπιστήμια. Ίσως θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν κάποιες προδιαγραφές, κάποιους δείκτες που θα μπορούσαμε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να κάνουμε μια κάποια σύγκριση. Ευχαριστώ κυρία Χάνιμπαλ, εκ νέου. Ναι, σα ευχαριστώ που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Λίγα στοιχεία να αναφέρω για το που θα επικεντρωθεί οι σοσιαλδημοκράτες. Πολλά ακούσαμε, αλλά θεωρώ ότι ίσως ο εισηγητής θα ήθελε να τα ξανακούσει. Η κοινωνική ε, συνοχή και ενσωμάταση και η προστασία των ε, μειονεκτούντων ομάδων. Πολύ σημαντικά στοιχεία και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να δράσουμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή Προστασία με νέα αξία και εδώ νομίζω ότι υπάρχει και η ενθάρρυνση και η υποστήριξη του αθλητισμού θα μπορούσαν να κάνει μεγάλη διαφορά, ιδιαίτερα σε μειονεκτούσες ε, κοινωνίες. Σύμφωνο ότι για τον ντόπινγκ θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταπολεμήσουμε στον αθλητισμό και επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της βίας. Αποτελούν τεράστιο θέμα και φυσικά υπάρχει και κάτι άλλο που αναφέρεται, το όλο θέμα της υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά το θέμα της υγείας και συνδρομή του αθλητισμού σε αυτήν. Γιατί συχνά οι νέοι ασκούν αθλητισμό όταν είναι νεαροί και μετά αυτό τους ε, έχει αποτελέσματα σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Επίσης να υποστηρίξω αυτά που ακούσαμε και για το στοιχηματισμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα σας υποστηρίξουμε απόλυτα. Και επίσης έγινε γραπτή δήλωση από τα μέλη της Επιτροπής αυτή για το θέμα αυτό. Αυτά τα βασικά στοιχεία που ήθελα να αναφέρω, το ξέρω ότι καλύπτω τα πιο πολλά εξ αυτών, απλά να αναφέρω ότι σας υποστηρίζουμε σε όλα αυτά. Εκτός μικροφώνη, πρόεδρος. Δεν μου αρέσει να διαβάζει κανείς ε, επιστολές συναδέλφων. Δεν έχει νόημα να μας λέτε τι θα έλεγε κάποιος αν θα ήταν εδώ. Πέντε λεπτά, Σαντιάγκο, όχι παραπάνω. Ας πούμε, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Έχω τα προβλήματά μου σήμερα γιατί βιάζομαι από ό,τι βλέπετε. Ζητώ συγγνώμη. Ποτέ δεν συμπεριφέρομαι έτσι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. να απαντήσω και εγώ στις πολλές παρατηρήσεις που ακούστηκαν από τον κύριο Φίσα και από τους άλλους ευρωβουλευτές όσον αφορά το σχέδιο δράσης ε, της ε, 23 Τετάρτης Μαΐου, το οποίο έκριναν οι Υπουργοί είναι σίγουρα η σημαντικότερη εξέλιξη που είχαμε στον αθλητισμό του τελευταίου μήνε. Αυτό το σχέδιο δράση το Συμβούλιο χαιρετίζει την ακίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ιανουαρίου και εγκρίνει τα θέματα τα οποία θίγονται στο κείμενο αυτό, θέτει όμω και κάποιε σαφεί προτεραιότητε για τα επόμενα τρία χρόνια. Προκειμένου να ασχοληθούμε με τι προτεραιότητε αυτέ, δημιουργούνται έξι θεματικές ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα επικεντρωνώνται σε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες περιγράφονται στο ψήφισμα αυτό. Θα ήθελα να αφαιρθώ σύντομα στις πιο σημαντικές από αυτές γιατί θα δείτε ουσιαστικά ότι κατοπτρίζουν τη συζήτηση των τελευταίων 25 λεπτών. Η πρώτη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα έχει να κάνει με το anti-doping που θα δημιουργήσει ένα νέο κείμενο για την αναθεώρηση του φυσταμένου κειμένου. Το δεύτερο, η δεύτερη ομάδα θα έχει να κάνει με τη χρηστή διακυβέρνηση. Έχει ως στόχο να δημιουργήσει συνθήκες διαφάνειας για την οικότητα αθλητισμό και να καταπολεμήσει το φαινόμενο των στημένων παιχνιδιών και το φαινόμενο των παρατυπιών όσον αφορά τις μεταγραφές. Όσον αφορά στη συνέχεια τους μάνατζερ, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς διοργανώσαμε μία συνδιάσκεψη με όλους τους εμπλεκομένους θα οργανώσουμε, συγχωρείτε, μια συνδιάσκεψη και ελπίζουμε αυτό να συνάδει κάπω και με την περίοδο εκείνη που θα γίνει μια πρόταση από τη FIFA και ουσιαστικά να καταφέρουμε να συμμορφωθούμε κάπω και με το δικό του το χρονοδιάγραμμα. Η επόμενη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα έχει να κάνει με την κατάρτιση και τον αθλητισμό. Θα δημιουργηθούν εδώ πέρα κάποιε κατευθυντήρε γραμμέ όσον αφορά την κατάρτιση στον αθλητισμό την καρδιδρομία στον αθλητισμό. Η άλλη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα έχει να κάνει με κάποιες συστάσεις του Συμβουλίου όσον αφορά την εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού, αθλητικές στατιστικές θα είναι η άλλη ομάδα εμπειρογνωμόνων και η τελευταία ομάδα εμπειρογνωμόνων θα έχει να κάνει με την χρηματοδότηση του αθλητισμού και την βιωσιμότητα προκειμένου να δημιουργηθούν κάποιοι μηχανισμοί υποστήριξη του αθλητισμού σαν αυτούς του οποίους πρότεινε η κυρία Μακλάρκιν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμφωνεί με τις προτάσεις αυτές που κάνει το Συμβούλιο. Πρόκειται σαφώς για κάποιες προτεραιότητες που θα εμπλουτίσουν τα μελλοντικά σχέδια ε, δράσης. Θέλουμε λοιπόν οι ομάδες αυτές εμπειρογνωμόνων, οι έξι που θα δημιουργηθούν, να είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές. Παράλληλα θα ξεκινήσουμε κι εμείς κάποιες ε, μελέτες που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την εργασία αυτών των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Μια, μια μελέτη που θα έχει να κάνει με, τη... με τα στημένα παιχνίδια, μια άλλη που θα έχει να κάνει με τις μεταγραφές, μια άλλη, ομάδα που θα έχει... μια άλλη μελέτη που θα έχει να κάνει με την ε, ε, ενίσχυση του αθλητισμού. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ε, να θα έχουμε και μια μελέτη όσον αφορά την χρηματοδότηση των ε, αθλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Επίσης προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τις προπαρασκευαστικές δράσεις του 2009-2010. Την αποτίμηση αυτή θα την έχουμε τις επόμενες εβδομάδες και θα τροφοδοτήσει και αυτή τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πολιετές ε, προγραμματικό πλαίσιο και θα μπορούσαν ουσιαστικά όλα αυτά να αποτελέσουν τμήμα ενός ξεχωριστού προγράμματος για τον αθλητισμό, στο οποίο αναφέρθηκε η Επίτροπος Βασιλείου πριν από λίγο και αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά και στις προτάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διαφορετικά ταμεία και νομίζω ότι έτσι απαντάω και στην αδελφό σας που έθεσε σχετικό ερώτημα. Ευχαριστούμε, Σαντιάγκο, πολύ σύντομα. Ε, Ευχαριστώ, θα κάνω ό,τι μπορώ, κύριε Πρόεδρε. Να πω πρώτα απ' όλα ότι συντάσσοντας την έκθεση αυτή απογοητεύτηκα λίγο γιατί είμαι στο τέταρτο προσχέδιο, έχω συναντηθεί με πάρα πολλούς ανθρώπους, έχω λάβει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όχι ότι ε, πρέπει να λάβω υπόψη όλα όσα μου έχουν πει, απλά συλλέγω και συγκεντρώνω πληροφορίες και για να το κάνω αυτό καλύτερα θεώρησα πρέπει να μιλήσω με κάθε είδους οργανώσεις, σε διάφορα άτομα, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο ούτε χώρο για την έκθεσή μου και πρέπει να δούμε και τις τροπολογίες είτε τις δικές μου είτε των άλλων ε, συναδέλφων. Δυστυχώς δεν μπορούν όλα να τα, δεν μπορώ όλα να τα περιλάβω στην αρχική έκθεση. Τηλεγραφικά μπορώ να πω αυτά πάντως. Τώρα, παντώντας ε, στο συνεδράς, πρώτα απ' όλα στον Ιβο Μπέλετ. Σίγουρα το διάβλητο είναι πολύ σημαντικό για τους ε, αγώνες και έχω αφιερώσει ειδική παράγραφο Μπορώ και να σας τη διαβάσω, αλλά δεν ξέρω αν χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικό. Προσπάθησα να αποφύγω να μιλήσω για UEFA, FIFA, να βάζω ονόματα και επώνυμα, να κατονομάζω. να μην ήταν ό,τι καλύτερο για την έκθεση. Αλλά βασίστηκα σε γενικές αρχές που πρέπει να τις σέβονται όλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να εισαγάγει ειδική τροπολογία γι' αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι είχα διάλογο μαζί τους, μίλησα μαζί τους και μου έκανα να καταλάβω και κάποια πράγματα που αρχικά εγώ ε, δεν ήξερα, είχα άλλη εικόνα. Και κάποια από τα αιτήματα τα έλαβε υπόψη. Παραδείγματο χάρη για το καθεστώ των αθλητικών συλλόγων, των αθλητικών σωματείων, το είπα. Για τα μικρά σωματεία κυρίω πρέπει να μιλήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικέ δυσκολίε χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και φυσικά διακυβέρνηση, που το είπαμε και αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα η ιδιαιτερότητα του κόσμου του αθλητισμού νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει. Αλλά παραλαμβάνω, πρέπει να το μελετούμε κατά περίπτωση και πρέπει να υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα, κάποια αντισταθμίσματα που θα πει διαφάνεια πλήρη και δημοκρατία πλήρη. Αλλιώ γιατί να δώσουμε πλεονεκτήματα, γιατί να δώσουμε προνόμια στον αθλητισμό. Στην κυρία Χάνιμπολ θέλω να πω ότι κοινωνική ένταξη είναι κάτι το οποίο σχολίασα ήδη. Θεωρώ ότι είναι σημαντική, θεμελιώδης. Ο αθλητισμός είναι κατά την άποψή μου η ιδανική μέθοδος για την κοινωνική ένταξη πολλών κοινωνικών ομάδων και εντός και εκτός Ευρώπης. Επίσης, μίλησαμε για την υγεία, το σχολίασα και το είπα και στην ίδια την Επίτροπο πριν. Θα έλεγα ότι όχι μόνο για την υγεία των νέων, αλλά και για τον ε, ηλικιωμένο, είναι πολύ σημαντικός αθλητισμό για τον ε, κύριο Τέρι, ο οποίος σχολίασε τα στημένα παιχνίδια. Φυσικά και είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και εγώ είπα ότι προτείνω να υπάρχει, ε, μια, να υπάρχει ποινικό αδίκημα για το στήσιμο των αγώνων. 3,65% του ΑΕΠ και το 5,4% του, ε, της απασχόλησης ε, είναι στοιχεία τα οποία έχω για τον αθλητισμό. Πόσο σημαντικός είναι η ε, κυρία ε, Μπασκούτ ε, που μου ζήτησε να της δώσω κάποιες εξηγήσεις. Δεν είμαι κατά του ΤΑΣ. Το ΤΑΣ είναι στην... Το ΚΑΣ συγκεκριμένα το λέμε στα ελληνικά. Αυτό το δικαστήριο είναι στην Γενέβη και έχει και στην Αυστραλία και στις ΙΠΑ μια αντιπροσωπεία, ένα παράρτημα. Γιατί να μην έχει και στην Ευρώπη, αυτό λέω. Το, νομικό, το ελβετικό νομικό σύστημα είναι τελείως διαφορετικό από το ευρωπαϊκό. Τι γίνεται λοιπόν, πολλοί αθλητές πηγαίνουν στο ΚΑΣ, δεν πείθονται από το ΚΑΣ και πάνε στην, ε, στα δικαστήρια ε, τα κανονικά της ε, χώρας τους. Αν το ΚΑΣ είχε μεγαλύτερη ξοπιστία στην Ευρώπη και βασιζόταν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα μπορούσαμε να αποφύγουμε ε, την προσφυγή στα εθνικά τακτικά δικαστήρια. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και να το μελετήσουμε. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των ε, χούλιγκαν και τι απαγορεύσει, νομίζω ότι κάθε κράτο πρέπει να θεσπίσει ένα κατάλογο των βίαιων, ανεπιθύμητων οπαδών, αυτών που δείχνουν ρατσιστική συμπεριφορά και πιστεύω ότι επίση πρέπει να γίνει μια κοινή λίστα που θα την έχουν στη θέση του όλα τα κράτη-μέλη. Και σε αυτού του χούλιγκαν δεν θα επιτρέπεται η σύσοδο στου αγωνιστικού χώρου, στα συμμετοχή του σε διάφορε αθλητικέ διοργανώσει. Μια πρόταση είναι αυτό, γιατί FIFA τα πάμε. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο Πιόρ Μπόρι, νομίζω ότι είναι προφανέ η χρηματοδότηση. Πολύ σημαντικό. Μία από τι προτάσει που θα κάνω είναι τα ευρωπαϊκά διαθροτικά ταμεία να ε, χρησιμοποιούνται και για τον αθλητισμό. Που αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Για την παιδεία ισχύει, όχι για τον αθλητισμό. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πράγματι, ακόμα καλύτερα αν χρηματοδοτήσει τον αθλητισμό. Για την Emma Μακλάρκιν και τη χρηματοδότηση, το συζητήσαμε νομίζω αυτό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω πάντω ότι υπάρχει και ένα θέμα που πρέπει να είναι σαφέ για όλου μα Και κυρίω γιατί εγώ σέβομαι την αυτονομία των ομοσπονδιών, αλλά και τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των κρατών μελών. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση. Θέλουμε να στηρίξουμε τον ε, ερασιτεχνικό, τον μαζικό αθλητισμό, αλλά αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά των κρατών μελών ή και των περιφερειών σε πολλέ περιπτώσει. Μπορούμε λοιπόν να δίνουμε συμβουλές, να επιμένουμε ότι είναι ένα θέμα πρωταρχική σημασίας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε εμεί από εδώ μέτρα, γιατί ουσιαστικά παραβιάζουμε με τον τρόπο αυτό την αρχή της επικουρικότητα. Δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε πάνω σε θέματα που δεν είναι δική μα αρμοδιότητα. Επαναλαμβάνω δε ότι σέβομαι γιατί εγώ προέρχομαι από τον κόσμο των ομοσπονδιών, εγώ σέβομαι ε, απόλυτα την αυτονομία των ομοσπονδιών, αλλά πρέπει να υπάρχει αντιπροσώπευση και διαφάνεια ό,τι αφορά τη σημαία. Υπόδειξη, δεν θέλω να επιβάλλω τίποτα. Για τον Μάρκο Σκουρία να πω, μίλησε για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του Αθλητισμού και εγώ πιστεύω σε αυτό και λειτουργεί καλά νομίζω ο θεσμός και θα πρέπει να το στηρίξουμε με δύο προϋποθέσεις. Θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση έστω και μικρή από την Κομισιόν αφενός και αφετέρου θα πρέπει να υπάρχει θα έλεγα μια εποπτεία, ένα έλεγχο του πώς γίνονται τα πράγματα. Πάντως πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό. Επίσης για τις γυναίκες. Οι γυναίκες και ο αθλητισμός είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Στον τρίτο κόσμο σίγουρα θα μπορούσε να, να συνεισφέρει στο να συναυθούν συμφωνίες ε, σε σχέση και με τη θέση την κατάσταση της γυναίκας. Εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ να προτείνω πολλά. Ε, δεν μ' αρέσουν οι ποσοστώσει, δεν πιστεύω στις ποσοστώσει. Φυσικά και θέλω τη μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Όχι, δεν το είπε κανεί, λέει εκτό ε, μικροφώνου σχόλιο ο κύριο Φίσα. Δεν, είπαμε ότι, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τόσε γυναίκε σε μια ομοσπονδία. Απλά λέω ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ε, συμμετοχή. Και τελικό, τελευταίο σχόλιο. Χαίρομαι που η Κομισιόν και το Συμβούλιο φαίνεται να υπέρ ε, μιας ε, πολιτικής, ενός προγράμματος για τον αθλητισμό. Αυτό είναι κοινοτομία. Και σε αυτές τις επιτροπές που θα δημιουργηθούν, καλό θα ήταν να εκπροσωπείτε το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Σαντιάκο. Σας ευχαριστούμε πολύ για το μεγάλο όγκο δουλειά και για την ε, πολυμορφία της έκθεσής σου. Νομίζω ότι όλα αυτά θα τα καταφέρεις εντός των ε, προδιαγεγραμμένων προθεσμιών. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να τα αποφασίσουμε αυτά ούτως. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούνται πάρα πολλά ε, στοιχεία, πολλά υποσχόμενα. Δεν το πιστεύουμε αυτό πάντα εξ αρχής, αλλά προφανώς ε, ήταν πιο σοβαρά τα σχόλια που ακούσαμε και μας είπε η Επίτροπο σήμερα ότι θα προκύψει τελικά ένα πρόγραμμα. Θα ήταν καλό να θέσετε λοιπόν τη σχετική βάση. Τον Ιούλιο θα παρουσιάσετε την έκθεση στον Σαντιάγκο και πότε θα ψηφίσουμε. Τον Οκτώβριο. Τέλεια. Έχουμε λοιπόν χρόνο μπροστά μας. Θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό στην Επιτροπή. Και τώρα πέρα στη συνεδρίασης, αύριο το πρωί στις 9 τα ξαναλέμε, όλοι όσοι δεν ε, έχουν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση των συντονιστών παρακαλώ να βγουν γρήγορα γρήγορα από την αίθουσα για να ξεκινήσουμε κατευθείαν τη συνεδρίαση των συντονιστών.